Good afternoon. Καλησπέρα σας αγαπητοί συνάδελφοι. Καλώς ήρθατε και πάλι. Θα ήθελα να καλωσορίσω θερμότατα την ομιγυρή και κυρίως όλους τους βουλευτές που έχουν έρθει και από άλλα μέρη της Ευρώπης και της Ασίας. Το πάνελ μας θα συζητήσει για τις κλιματικές αλλαγές, τις ε, περιβαλλοντικές προκλήσεις και τον αντίκτυπό του στην οικονομία. Γνωρίζω ότι μερικοί για να έρθετε χρειάστηκε να ταξιδέψετε πολλές ώρες και ελπίζω ε, να πιάσει τόπο το ταξίδι σας, γιατί ε, βλέπουμε και στην Ασία αλλά και στην Ευρώπη μερικές πολύ ριζικές αλλαγές στο κλίμα. Και η κατάσταση αυτή χρήζει έκτακτης και πολυμερούς συνεργασίας. Και γι' αυτό σε ευχαριστώ θερμά για την παρουσία σας εδώ σήμερα, γιατί έτσι θα συμβάλλουμε, μόνο έτσι θα καταφέρουμε να σημειώσουμε πρόοδο, αν συνεργαστούμε και προτείνουμε ιδέες για να ξεπεράσουμε όλες τις προκλήσεις. Κάτι που προϋποθέτει ε, μεγαλύτερη ενίσχυση και των κοινοβουλευτικών πλατφορμών και φόρουμ και με την σύσφυξη των κοινοβουλευτικών σχέσεων ε, μεταξύ Ασίας και Ευρώπης. Και ο λόγος που βρισκόμαστε εδώ είναι γιατί αναγνωρίζουμε πως οι κλιματικές αλλαγές δεν γνωρίζουν σύνορα. Δεν γνωρίζουν η η η μισφαίρια. Και επίσης επηρεάζουν δραστικά την καθημερινότητα των συμπολιτών μας αλλά και την οικονομία μας. Και μάλιστα το καλοκαίρι που μας πέρασε είδαμε άνευ προηγουμένου βροχοπτώσεις με πλημμύρες στην Ινδία, στη, στο Μπαγκλαντές και ταυτόχρονα είχαμε ένα καύσωνα στην Ευρώπη με πυρκαγιές στην Ελλάδα και τη Σουηδία και τυφώνες που γίνονται όλο και δρυμύτεροι και πιο καταστροφικοί κάτι που επηρεάζει ιδιαίτερα και την παραγωγή τροφίμων στην Ασία. Θα πρέπει λοιπόν να κάνουμε τη μετάβαση σε πιο σε οικονομίες που θα έχουν χαμηλότερες εκπομπές άνθρακα και θα πρέπει να δούμε πώς θα υιοθετήσουμε μια στρατηγική που θα συνδέει την Ευρώπη και την Ασία. Και μάλιστα η προσέγγιση μας στην συνδεσιμότητα ε, δίνει έμφαση στην βιωσιμότητα σε πολλά επίπεδα, όχι μόνο σε οικονομικό και φυσικό επίπεδο, αλλά και σε κοινωνικό και πάνω απ' όλα σε περιβαλλοντικό επίπεδο. Θα πρέπει λοιπόν να συνεργαστούμε ώστε να μετατρέψουμε τις σημερινές προκλήσεις σε ευκαιρίες. Η περιβαλλοντική προστασία μπορεί να συμβάλλει στην οικονομική ανάπτυξη και στην κοινωνική ευμάρεια. Και γι' αυτό υιοθετήσαμε στην Ευρωπαϊκή Ένωση ένα φιλόδοξο πακέτο για την κυκλική οικονομία που θα συμβάλλει στην ε, ενθάρρυνση της ε, ευρωπαϊκής οικονομίας σε μια κυκλική οικονομία, με χαμηλότερε εκπομπέ άνθρακα και με δημιουργία νέων θέσεων απασχόληση. Θέλουμε να μειώσουμε τα απόβλητα, να αυξήσουμε την ανακύκλωση και την επαναχρησιμοποίηση των υλικών. Κάτι που θα ωφελήσει και το περιβάλλον και την οικονομία. Η Ευρωπαϊκή Ένωση λοιπόν προσπαθεί να ενισχύσει τη συνεργασία και με την Ασία στον τομέα της περιβαλλοντικής πολιτικής. Και χαίρομαι ιδιαίτερος που έχουμε ένα πακέτο με τόσο κορυφαίους εμπειρογνώμονες που θα δώσουν τροφή στη συζήτηση και ελπίζω σε τη συζήτηση που θα ακολουθήσει να συμμετέχετε ενεργά όσο περισσότερο γίνεται. Εγώ θα ήθελα να κάνω κάποιες διαδικαστικές ε, παρατηρήσεις πριν σας παρουσιάσω το πάνελ και δώσω τις κοιτάλες στον Συμπρόεδρο. Να σας υπενθυμίσω ότι έχουμε διερμηνία σε όλες τις γλώσσες Ευρωπαϊκής Ένωσης με εξαίρεση τα Ιρλανδικά και Ελτικά αλλά έχουμε και άλλες γλώσσες Ρωσικά στο κανάλι 27 Χμέρ στο 25 Βιετναμέζικα στο κανάλι 26 και Μογγολικά στο κανάλι 29 όπως σας είπα θα ακούσουμε πρώτα τους ε, έμπειρογνώμονές μας και θα ακολουθήσει γύρω σε ερωταπαντήσεων. Και τα τρία πάνελ αύριο το πρωί θα μας ενημερώσουν για τα πεπραγμένα τους. Οπότε θα πρέπει να ορίσουμε έναν εισηγητή που θα παρουσιάσει αύριο τα αποτελέσματα της σημερινής μας συζήτησης. Και δεν ξέρω ποιος θα ήθελε από την Ομίγυρα να λάβει αυτό το ρόλο του εισηγητού. Παρακαλώ. Υπάρχει εθελοντής ή να το αφήσουμε για αργότερα. Καλό θα ήταν όμως από τώρα να γνωρίζουμε ποιος ε, θα είναι ο εισηγητής μας και ποιος θα ενημερώσει αύριο την Ολομέλεια για τις εργασίες της ομάδας μας. Υπάρχει κάποιος εθελοντής, εθελοντές για την αυριανή ενημέρωση. Το όνομά σας παρακαλώ. Φραντσέσκο Τζάκοβό από την Ιταλική Γερουσία. Σας ευχαριστούμε κύριε Γερουσιαστά. Οπότε, ίσως στο τέλος θα μπορούσατε να κάνετε μια σύντομη ανακεφαλαίωση και να μας πείτε τι θα πείτε αύριο στην Ολομέλεια. Με ιδιαίτερη χαρά τώρα θα δώσω τη σκητάλη ε, στον συμπρόεδρο καθηγητή Γιουέν από το Πανεπιστήμιο του Τσίγουα που είναι ε, και αντιπρόεδρος του Πανεπιστημιακού Συμβουλίου. Έχετε το λόγο κύριε καθηγητά. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Είμαι από την Κίνα. Δεν έχουμε φέρει διερμηνέα Κινέζο, Κινέζικη και γι' αυτό θα προσπαθήσω να μιλήσω αγγλικά, αν και τα αγγλικά μου τα έμαθα στην Κίνα. Οπότε ζητώ την επίοικιά σας. Θα ήθελα να σας παρουσιάσω τους δύο κεντρικούς μας ομιλητές στο δικό μας πάνελ. Ο πρώτος είναι ο κύριος Κόλεν Άλεν που είναι πρόεδρος της Επιτροπής Α, συγγνώμη λέει ο ομιλητής. Κυρία Πρόεδρε, έχω ετοιμάσει ένα σύντομο μήνυμα και η συμπρόεδρος μου λέει να το διαβάσω πρώτα αυτό. Οπότε πρώτα θα σας διαβάσω το σύντομο μήνυμα και μετά θα σας παρουσιάσω τους κεντρικούς μας ομιλητές. Νιώθω ιδιαίτερη χαρά και μεγάλο προνόμιο που μου δίνει τη ευκαιρία να σας παρουσιάσω κάποιες ιδέες εδώ. Οι κλιματικές αλλαγές αποτελεί κοινή πρόκληση ολόκληρης της ανθρωπότητας είναι μια πρόκληση που αναγκάζει ολόκληρη την ανθρωπότητα να ε, δράσει ώστε να αντιμετωπίσει τις κλιματικές αλλαγές ε, ε, για το παγκόσμιο περιβάλλον. Σε ό,τι αφορά το κλίμα και το περιβάλλον, θα πρέπει να εθετήσουμε μια ολοκληρωμένη ολιστική προσέγγιση που θα περιλαμβάνει και την οικονομική πτυχή και την κοινωνική πτυχή αλλά και πολλούς άλλους παράγοντες ταυτόχρονα. Γιατί δεν είναι σωστό να επιδιώκουμε μόνο την ικανοποίηση οικονομικών συμφερόντων ε, και να θυσιάζουμε το περιβάλλον μας στο βωμό της οικονομίας. Γιατί πολλοί συμπολίτε μας έχουν ε, εύλογη ανάγκη επιβίωσης ε, και χρήζουν προστασίας, το ίδιο και το περιβάλλον. Και γι' αυτό, για να αντιμετωπίσουμε τις κλιματικές και περιβαλλοντικές προκλήσεις, θα πρέπει πρώτα να αντιληφθούμε σωστά τις εξελίξεις στην οικολογία και θα πρέπει να τηρήσουμε τους νόμους της φύσεως αποφεύγοντας τη διάπραξη λαθών όταν προσπαθούμε να χρησιμοποιήσουμε και να εκμεταλλευτούμε τη φύση. Επίσης, θα πρέπει να αναλάβουμε από κοινού τις ευθύνες μας και Επίσης, να λάβουμε υπόψη και τις διάφορες εθνικές πραγματικότητες, τις ικανότητες που έχουν τα διάφορα κράτη και τις ανάγκες των αναπτυσσόμενων χωρών. Και μάλιστα η Κίνα θεωρεί ότι υπάρχει μεγάλος συνδεσμός μεταξύ της οικολογίας του περιβάλλοντος, ε, της οικονομίας και του κοινωνικού περιβάλλοντος. Και Γι' αυτό θέλουμε να δημιουργήσουμε ένα νέο αναπτυξιακό μοντέλο που θα διέπεται από την ιδέα της προσαρμογής ε, στη φύση και της προστασίας της φύσης. Και από το 2005 μέχρι το 2015 το 5,1% της ε, ενεργειακής κατανάλωσης ε, που έχει αυξηθεί συνοδεύτηκε με 9,5% αύξηση ετησίως της οικονομικής μας ανάπτυξης. Και μάλιστα η οικονομική ανάπτυξη και οι εκπομπές ε, διοξιδίου του άνθρακα συνδέονται όλο και λιγότερο μεταξύ τους. Και το παράδειγμα της Κίνας έχει αποδείξει ότι η καταπολέμηση των κλιματικών αλλαγών και η εξασφάλιση της περιβαλλοντικής προστασίας ε, ε, μπορούν να συμβαδίσουν με την οικονομική ανάπτυξη. Και μάλιστα στο μέλλον η Κίνα θα εξακολουθήσει να είναι δεσμευμένη στο, στο μονοπάτι της οικονομίας χαμηλών εκπομπών άνθρακα και προσβλέπει σε μια πράσινη οικονομία απαλλαγμένη από τον άνθρακα και μια κυκλική οικονομία με την ενίσχυση της οικονόμησης ενέργειας και της περιβαλλοντικής προστασίας. Θέλουμε ένα ενεργειακό σύστημα που θα είναι καθαρό, θα έχει χαμηλές εκπομπές άνθρακα και επίσης θα προωθήσουμε ένα βιωτικό μοντέλο οικολογικό. Τώρα επανέρχομαι στα παγκόσμια περιβαλλοντικά ζητήματα που είναι αδύνατο να αντιμετωπιστούν χωρίς διεθνή συνεργασία. Είναι επιτακτική ανάγκη όλες οι χώρες, οι κοινωνικέ ομάδε, αλλά και οι ιδιώτε, να συντονίσουν τι προσπάθειε του. Η Κίνα πρότεινε τη δημιουργία μιας κοινότητας με κοινό μέλλον, που είναι η ολόκληρη ανθρωπότητα και θα πρέπει να αξιοποιήσουμε τις κοινέ μας γνώσεις για να αντιμετωπίσουμε κοινά προβλήματα όπως είναι οι κλιματικές αλλαγές και το περιβάλλον. Θα πρέπει να ξεπεράσουμε ε, κάποιες ε, παλιές ε, ιδεολογίες όπως της, του ωφελημισμού και της ανάγκης να βγούμε όλοι κερδισμένοι, γιατί κάτι τέτοιο θα αποβεί βάρος μας. Μόνο προωθώντας την ιδέα μιας κοινότητας με κοινό μέλλον μπορούμε όλοι να ανασκομποθούμε και να ενώσουμε τις προσπάθειές μας για να εξασφαλίσουμε το κοινό μας μέλλον. Και μάλιστα στο μέλλον, έχοντας μια κοινότητα με μέλλον για όλη την ανθρωπότητα, η Κίνα θα διαδραματίσει ενεργά το ρόλο της σε μια παγκόσμια κλιματική και περιβαλλοντική διακυβέρνηση και θα συνεισφέρει στην προστασία της επικράτειάς της και για τις μελλοντικές γενιές. Αυτό είναι το μήνυμά μου, κυρία Πρόεδρε, και αυτές ήταν οι ιδέες της κινέζικης αντιπροσωπείας. Και τώρα θα ήθελα να σας παρουσιάσω τους κεντρικούς μας ομιλητές. Ο πρώτος ομιλητής μας Ο πρώτος ομιλητής μας είναι ομιλήτρια. Είναι η κυρία Λίντι Νάκπιλ, συντονίστρια στο κίνημα των ασιατικών λαών για το χρέος και την ανάπτυξη. Ευχαριστώ πολύ. Λέγομαι την Νάκπιλ, είμαι από τις Φιλιππίνες και εργάζομαι με μια σειρά κινημάτων της κοινωνίας των πολιτών στην Ασία για το θέμα της ε, αλλαγής του κλίματος. Σας ευχαριστώ που μας δώσατε την ευκαιρία να μιλήσουμε στο φόρουμ σας. Ο αντίκτυπο της κλιματική αλλαγή ε, στην οικονομία ήδη είναι τεράστιο, ε, ιδίω για τις πιο ευπαθείς χώρες και πολλέ από αυτέ βρίσκονται στην Ασία. Θα είναι μαζικό και θα κλιμακωθεί πριν να σταματήσουμε, να μπορέσουμε να σταματήσουμε την υπερθέμαση του πλανήτη και να σταθεροποιήσουμε το κλίμα. Θέλω να τονίσω τρεις τομείς που για μας είναι επίγοντες. Ε, αυτό δεν σημαίνει ότι δεν υπάρχουν ε, άλλοι επίγοντες τομείς, αλλά σε μία σύντομη παρουσίαση νομίζω ότι πρέπει να αναφερθώ κυρίως σε αυτούς τους τρεις που είναι πιο σημαντικοί. Καταρχήν ε, για τα τρόφιμα και την παραγωγή των τροφίμων. Η κλιματική αλλαγή και θα έχει μεγάλο αντίκτυπο στην ικανότητά μας να παράγουμε τρόφιμα, να έχουμε πρόσβαση στα τρόφιμα και ε, στο είδος των τροφίμων που μπορούμε να καταναλώσουμε. Η κλιματική αλλαγή ε, κλιμακώνει ήδη σοβαρές ε, κρίσεις τροφίμων και πείνα και λοιμούς σε πολλά μέρη του κόσμου. Ε, έχουμε ε, πολλές, ε, πολλές συχνά φαινόμενα όπως ξηρασίες, τυφώνες, τη γη που γίνεται αλμυρή, έχουμε καιρικά φαινόμενα, απρόβλεπτα, όλα αυτά θα έχουν αντίκτυπο στη γεωργία. Η υπερθέρμανση των ωκεανών και η οξύνηση των ωκεανών, η αλλαγή Τη κίνησης ε, του νερού των ωκεανών, των υδάτων των ωκεανών, αυτά έχουν μεγάλο αντίκτυπο ε, στα αλλιεύματα, στο μέγεθος ε, των ψαριών και στα μεταναστευτικά μοντέλα των ψαριών. Θέλουμε να τονίσουμε ότι ένα σημαντικό μέρος του παγκοσμίου πληθυσμού και εμείς από τις Φιλιππίνες εξαρτόμαστε από τα ψάρια ως την κύρια πηγή πρωτεΐνης. Επομένως είναι κατεπήγον στο θέμα της παραγωγής των τροφίμων όχι απλώς ε, να σκεφτούμε ε, πώς θα οικονομήσουμε ανθεκτικότητα σε ό,τι αφορά τη γεωργία και την προστασία των υδάτινων πόρων, αλλά να ε, αναθεωρήσουμε και τη χρήση της γης και το να έχουμε προτεραιότητες για την παραγωγή του τροφίμων. Εμείς στο Κοινοβούλιο στις Φιλιππίνες έχουμε προωθήσει ένα νομοσχέδιο για να αλλάξει η χρήση της γης και η πολιτική της χρήσης της γης, λαμβάνοντας υπόψη την μεγάλη, το μεγάλο αντίκτυπο της κλιματικής αλλαγής στην παραγωγή των τροφίμων. Η δεύτερη μεγάλη σύσταση που έχουμε είναι ότι οι χώρες μας, κυρίως οι αναπτυσσόμενες χώρες, θα πρέπει να θέσουν σε προτεραιότητα την παραγωγή τροφίμων για εγχώρια κατανάλωση. Σε πολλές χώρες έχουμε την εξή πραγματικότητα. Η παραγωγή μας στη Γεωργία, παραδείγματος χάρη, ακόμη και για την αλληλευτική βιομηχανία ε, είναι ότι δίνεται προτεραιότητα στις εξαγωγές. Αυτό πρέπει να αλλάξει. Ένας άλλος ε, τομέας ε, μεγάλης ανησυχίας είναι το μέγεθος και η συχνότητα ζημιών επειδή έχουμε ακραία καιρικά φαινόμενα και μεγάλο αντίκτυπο της αλλαγής του κλίματος. Κανένα, αν έχουμε μάλλον ε, ανθεκτικότητα στις αλλαγέ, αυτές θα μπορέσουν οι λαοί μα να αντισταθούν ε, στις επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγή. Δυστυχώ, οι διεθνεί διαπραγματεύσεις δεν συζητούν το θέμα το οικονομικό ως μέρος ενός διεθνούς προγράμματος για την αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής και της απώλειας και των ζημιών. Αυτό εμποδίζει την ε, πιθανή αποτελεσματικότητα του Διεθνούς Μηχανισμού για την Απόλυα και τη ζημία στην οποία ε, συμφώνησε ε, το 2013 Σύνοδος των Ηνωμένων Εθνών. Μία άλλη σύσταση είναι ότι ε, θέλουμε να πείσουμε τους βουλευτές να χρησιμοποιήσουν την επιρροή τους για να προωθήσουν αυτά τα θέματα περαιτέρω στις διεθνείς διαπραγματεύσεις. Ο επόμενο τομέα που θέλω να τονίσω είναι οι οικονομικές επιπτώσεις ε, της μετατροπής των συστημάτων ενέργειας. Είναι σαφές και ε, στο, το, η έκθεση του EPCC για το στόχο ε, του 1,5 βαθμού Κελσίου θα ξεκαθαριστεί περαιτέρω γιατί το έγγραφο αυτό θα εκδοθεί σε, κάποιες σε δύο εβδομάδε. προκειμένου να έχουμε εμεί τη δυνατότητα να κρατήσουμε την, θερμο, την αύξηση θερμοκρασία κάτω από τον 1,5-2 βαθμής ε, θα πρέπει να πετύχουμε το συντομότερο δυνατόν ε, μέχρι το 2050 ενέργεια 100% από ανανεώσιμε πηγέ. Αυτό έχει βαθιά επίπτωση στα οικονομικά μα συστήματα έχουμε κάποιες εκκλήσεις να απευθύνουμε. Καταρχήν, οι εθνικές ε, εισφορές ε, θα πρέπει να αυξηθούν, θα πρέπει να είναι πιο φιλόδοξες. Έχουμε ένα τεράστιο κενό φιλοδοξίας μεταξύ της μείωσης των εκπομπών θεωρίου του θερμοκηπίου για τις οποίες έχουν δεσμευτεί οι κυβερνήσεις μας και την πραγματική απέτηση να διατηρήσουμε την αύξηση της ε, κάτω του 1,5 των 2 βαθμών. Οι δεσμεύσεις που έχουν γίνει ως μέρος της Συμφωνίας των Παρισίων θα μας οδηγήσουν σε αύξηση θερμοκρασίας κατά 3 βαθμούς Κελσίου και ήδη ε, ενώ έχει αυξηθεί η θερμοκρασία κατά ένα βαθμό, έχουμε δει ότι έχουμε ιδιαίτερα καταστροφικές επιπτώσεις, όχι μόνο στην οικονομία συνολικά, αλλά και στους ίδιους τους λαού και τις κοινότητες. Επιπρόσθετα, έκκληση είναι σε όλες τις χώρες να σκεφτούν να αυξήσουν τη φιλοδοξία τους, όμως αυτή η έκκληση απευθύνεται κυρίως στις αναπτυγμένες, στις πλούσιες χώρες, καθώς οι δεσμεύσεις τους ουσιαστικά είναι πολύ μικρές ανάλογα με το μερίδιο που θα έπρεπε να έχουν στην καταπολέμηση κλιματικής αλλαγής. Το να πετύχουμε τους στόχους Παρισίου σημαίνει ότι πρέπει ε, να απομακρυνθούμε από τη χρήση ενέργειας απορρικτά καύσιμα, αλλά με έναν τρόπο που θα πρέπει να διασφαλίζει τη ε, δίκαιη μετάβαση. Η δίκαιη μετάβαση είναι μια έννοια πάρα πολύ σημαντική κυρίως ε, ως ελάχιστο θα πρέπει να έχουμε μια στρατηγική ε, να αντιμετωπίσουμε τη μετατόπιση ε, των εργαζομένων καθώς απομακρυνόμαστε από τη χρήση των πόρων και στη συνέχεια θα πρέπει να σταματήσουμε την περαιτέρω επέκταση του συστήματος ορεικτών καυσίμων και να έχουμε μια σταδιακή εξάλληψη προκειμένου να πετύχουμε τους στόχους μας. Και τέλος, για να επιλύσουμε την κλιματική κρίση θα πρέπει να επαναλάβουμε και να δώσουμε έμφαση στο ότι χρειάζεται βαθιά ε, τροποποίηση όχι μόνο των εθνικών οικονομιών αλλά και της παγκόσμιας οικονομίας στο σύνολό της. Θα πρέπει να στοχεύσουμε όχι μόνο να πετύχουμε οικονομικά συστήματα με χαμηλό άνθρακα ή μετά τον άνθρακα, αλλά επίσης στοχεύουμε στο να έχουμε οικονομικά συστήματα που να είναι δίκαια και ισότιμα. Σας ευχαριστώ. Ευχαριστούμε πολύ για την εξαιρετική σας αυτή παρέμβαση. Με χαρά να σας παρουσιάσω τον πρώτο βασικό μας ομιλητή, τον κύριο Κόλιν Άλεν, πρόεδρο της Επιτροπής Περιβάλλοντος της Ρουμανίας. Thank you, Mr. Chair. co-chairs. Ευχαριστώ. Αγαπητοί συμπρόεδροι, αγαπητοί συνάδελφοι, Αγαπητοί προσκεκλημένοι της ΑΣΕΠ 10, με χαρά μου βρίσκομαι εδώ για το πολύ σημαντικό αυτό ζήτημα για, την, για τον πλανήτη μας, την κλιματική αλλαγή. Και μιλώ σε ένα κοινό, κοινό το οποίο ε, είναι πολύ σημαντικό. Έχουμε την, ε, τα εργαλεία, αλλά χρειαζόμαστε και τη βούληση για να αντιμετωπίσουμε τα προβλήματα και η πλατφόρμα ASEP είναι εξαιρετική για αυτό το σκοπό. Η κλιματική αλλαγή αποτελεί τεράστια πρόκληση με μακροπρόθεσμες επιπτώσεις για την βιώσιμη ανάπτυξη και την ασφάλεια όλων των χωρών. Απειλεί να υποσκάψει την παγκόσμια σταθερότητα και ασφάλεια λόγω των επιπτώσεών της, όπως είναι η μαζική λοιμή, η έλλειψη νερού, η αναγκαστική μετάφραση ε, με, μετανάστευση, η διασπορά ασθενειών. Εκείνοι που αντιμετωπίζουν τους ε, σημαντικότερους κινδύνους βεβαίως είναι οι φτωχοί. Εκείνοι που έχουν τους λιγότερους πόρους για να αντιμετωπίσουν, παρόλο που εκείνοι φταίνε λιγότερο από όλου για την κρίση που αντιμετωπίζουμε. Ο πλανήτης μας αλλάζει. Έχουμε ρεκόρ καύσωνα ε, και υψηλών θερμοκρασιών τα τελευταία τρία χρόνια. Δερφορικά δεδομένα του Ιουνίου 2017 δείχνουν από το 1998 η υδρόγειος θερμαίνεται με διπλάσια ταχύτητα από ό,τι είχαν προβλέψει τότε οι επιστήμονες. Έχουμε πιο θερμούς και πιο όξινους ωκεανούς, έχουμε μείωση και τήξη των πάγων, έχουμε αύξηση της στάθμης των θαλασσών, έχουμε ακραία καιρικά φαινόμενα. Η προσαρμογή γίνεται λοιπόν βασικό στοιχείο και αναγκαίο στοιχείο για τον μετριασμό της κλιματικής αλλαγής από πλευράς μας. Και ενώ αυτός ο μετριασμός έχει, ε, έχει κατοχυρωθεί στους παγκόσμιους στόχους η προσαρμογή απαιτεί εθνική και τοπική αλλαγή σε κάθε χώρα ξεχωριστά. Αλλά δεν αρκεί, χρειάζεται να περισσότερο περισσότερα. Στο πλαίσιο λοιπόν τη συνάντηση κοινοβουλευτική εταιρική σχέσης τη Ευρώπη και τη Ασίας, αλλά και εν ώψη της προετοιμασίας της COP24 στην Πολωνία, αλλά και εν ώψη των συμπερασμάτων του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, είναι προφανές ότι η κλιματική αλλαγή απαιτεί ε, συγκεκριμένη και απτή δράση σε διεθνέ, εθνικό, περιφερειακό και τοπικό επίπεδο. Είναι καθήκον μας λοιπόν ως πολιτικών να προσδιορίσουμε την κλιματική αλλαγή ως ύψιστη προτεραιότητα και να θεσπίσουμε μέτρα τα οποία θα μας βοηθήσουν να επιτύχουμε τους στόχους μας. Δυστυχώς η κλιματική αλλαγή ε, θα είναι εδώ, ήρθε εδώ για να μείνει πολιτικοί που αγνοούν την κλιματική αλλαγή είναι πολιτικοί του παρελθόντος. Το περιβάλλον και το μέλλον του πλανήτη δεν μπορεί κανείς να τα αγνοήσει σε καμία πλέον απόφαση που θα παίρνετε από εδώ και στο εξή στις χώρες μας. Η ΑΣΕΠ εκπροσωπεί και αποτελεί το βασικότερο και το ιδανικότερο πλαίσιο και περιβάλλον για να συζητηθούν αυτά τα θέματα. Οι αποφάσεις μας για τις αλλαγές που θα εφαρμόσουμε είναι πολύ σημαντικές για τον ε, πλανήτη μας, καθώς οι χώρες ΑΣΕΜ αντιστοιχούν στο 60% του παγκόσμιου πληθυσμού. Έχουμε την εξουσία, τη δύναμη αλλά και τα εργαλεία για να επιτύχουμε τους στόχους, καθώς είμαστε σχεδόν το 2 τρίτα της παγκόσμιας οικονομίας και είμαστε ηγέτες στον τομέα της τεχνολογίας και της έρευνα. Και έχουμε βούληση να τα κάνουμε όλα αυτά, όπως αποδεικνύει και η διακήρυξη που θα υπογράψουμε αύριο. Και το πιο σημαντικό από όλα, ο καιρό είναι τώρα για να γίνουν όλα αυτά. Όταν ε, πριν από μερικά χρόνια τα αυτά που ε, συμβαίνουν σήμερα ε, ε αποτελούν σαν σενάρια επιστημονικής φαντασίας. Μπορούμε πραγματικά σήμερα πια να, να, να ταξιδέψουμε σε ολόκληρο τον κόσμο με ηλιακή ενέργεια και μόνο. Να ε, αυξήσουμε με αποτελεσματικότερη χρήση των υδάτινων πόρων τη γεωργία, την γεωργική μας παραγωγή. Όλα αυτά πλέον μας δίνουν τη δυνατότητα για να αντιμετωπίσουμε την παγκόσμια πρόκληση της κλιματικής αλλαγής. Και η Ρουμανία ε, επικυρώνοντας τη Συμφωνία των Παρισίων έχει αρθεί στο ύψος των περιστάσεων και των ευθυνών της και αποτελεί έναν από τους συγχρηματοδότες, ε, έναν από τους συνυπογράφοντες της, ε, του πρόσφατου ψηφίσματος της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΟΥ. Την επόμενη χρονιά, τον Απρίλιο του 2019, στο πλαίσιο της ε, Ρουμανικής Προεδρίας του Συμβουλίου, θα διοργανώσουμε και μια σχετική εκδήλωση που θα είναι αφιερωμένη στα προβλήματα και στους κινδύνους που προκαλεί η κλιματική αλλαγή αλλαγή και τα μέτρα που μπορούν να ληφθούν για την αντιμετώπιση αυτής. Ω αποτέλεσμα της COP24 που θα γίνει το Δεκέμβριο στο Κατοβίτσε της Πολωνία, είναι σημαντικό ε, να δοθεί συγκεκριμένος, ε, να, να θεσπιστούν συγκεκριμένα μέτρα που θα ληφθούν στο πλαίσιο των αποφάσεων των Παρισίων. Μετά το Κατεβίτσε θα γίνει και η εκδήλωση που σας ανέφερα στην ε, Ρουμανία υπό την Ρουμανική Προεδρία. Μας ενδιαφέρει πολύ να, αναλάβουμε, να λάβουμε τη σκητάλη από την Αυστρία που αυτή τη στιγμή βρίσκεται στην Προεδρία του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου και να συνεχιστούν οι διεθνείς συνομιλίες για την εξασφάλιση της σωστής υλοποίηση της Συμφωνίας των Παρισιών. Όλα αυτά τα μέτρα δείχνουν την προσήλωσή μας σε ένα βιώσιμο, υγιές και ασφαλές περιβάλλον για τον πλανήτη μας, για τις μελλοντικέ γενιές. Δεν είναι μόνο για το μέλλον μας, είναι ακόμη και η ίδια η ύπαρξη του μέλλοντος αυτή, του πλανήτη αυτό που διακυβεύεται. Και όπως είπα έχουμε τις αρμοδιότητες, την εξουσία, τη δύναμη, τους πόρους αλλά και τη βούληση για να τα κάνουμε όλα αυτά και ο καιρός πλέον είναι όριμος. Thank Σας ευχαριστώ. Κύριε Κόλιν Άλεν που ήταν ο πρώτος κεντρικός μας ομιλητής και τώρα με ιδιαίτερη χαρά θα καλέσω το δεύτερο μας κεντρικό ομιλητή Σέρι Σάμιν Κολτ από τον Μπαγκλαντές από τη μόνιμη επιτροπή Κοινοβουλευτική Επιτροπή του Μπαγκλαντές Αξιότιμοι συμπρόεδροι αξιότιμα μέλη του Εσέπ, κεντρικέ κύριε Κεντρική Μιλητά, Κόλιν Άλεν, αξιότιμοι συνάδελφοι. Χαίρομαι και με τιμά ιδιαίτερη συμμετοχή μου σε αυτή την 10η ΑΣΕΠ με θέμα την ε, οικονομία και το περιβάλλον. Και είναι ιδιαίτερο προνομιό μου που ως κεντρική ομιλήτρια θα σας παρουσιάσω κάποιες σκέψεις μου εδώ. Οι κλιματικές αλλαγές δημιουργούν τεράστιες απειλές στην οικονομική ευημερία και την ανάπτυξη και μάλιστα ε, ο διαδεδομένος και αν προηγουμένο ε, αντικτύπωση χτύπα κυρίως τους φτωχούς. Γι' αυτό χρειάζεται παγκόσμια δράση για να αντιμετωπίσουμε αυτές τις απελές χάρη σε παγκόσμια συνεργασία. Υπάρχει επιτακτική ανάγκη τέτοια συνεργασίας και στο πλαίσιο αυτό θα ήθελα να σας επισημάνω ότι το Μπαγκλαντές είναι από τις πιο ευάλωτες χώρες που έχουν πληγεί ιδιαίτερως από τις κλιματικές αλλαγές. Και παρόλο που είναι δύσκολο να κάνουμε ένα πλήρη απολογισμό του συνολικού αποτελέσματος των κλιματικών αλλαγών στην ευημερία και την οικονομία, λόγω των διαφόρων μεταβλητών και συνιστοσών σε τοπικό και εθνικό επίπεδο. Πάντω ε, μία μικρή αύξηση τη παγκόσμια θερμοκρασία έως και δύο βαθμούς ε, με βάση τα στοιχεία του 1990 θα οδηγήσουν ε, σε μείωση κατά μερικές ποσοστιαίες μονάδες το παγκόσμιο ΑΕΠ. Σε μερικές περιπτώσεις έχουμε κάποια μικρή αύξηση, αλλά σε λίγε περιπτώσεις μόνο. Αυτή ήταν η δήλωση του Σμιθ του 2001. Οπότε θα πρέπει να δούμε πώς επηρεάζει το το κλίμα και πώς επηρεάζουν οι κλιματικές αλλαγές στην οικονομία. Επίσης, πώς θα αποτιμήσουμε τις ακραίες καιρικέ συνθήκες που πλήττουν τη γεωργία και την παραγωγή τροφίμων και άλλες πτυχές κοινωνικο-οικονομικού χαρακτήρα που ε, δημιουργούν απόλυτες και αλλαγές. Επίσης, α, α, κλιματικές αλλαγές θα δημιουργήσουν κατά 5% μείωση του παγκόσμιου κατακεφαλήν εισόδημα. Επίσης, επηρεάζεται και το παγκόσμιο εμπόριο και όλο και περισσότεροι συνάνθρωποι μας οδηγούνται στην φτώχεια ε, Κυρίως η γεωργία πλήττεται, γιατί το κλίμα και η γεωργία είναι αλληλένδετα. Βέβαια, αναλύθηκαν πολλέ πολλές μεταβλητές για να εκτιμηθεί και να γίνει απολογισμός του αντικτύπου των κλιματικών αλλαγών στη γεωργία. Για παράδειγμα, 20 με 30% μείωση στην παραγωγή απορροκεπευτικών, λέει μια μελέτη του 1995. Επίσης, μια μελέτη του 2000 προτάθηκε ότι αύξηση ε, η παραγωγή ρυζιού στην ε, Ασία θα μειωθεί κατά 8% ε, κάτι που θα οδηγήσει σε μείωση του γεωργικού ΑΕΠ κατά 3,1% το χρόνο στην Ασία. Θα πρέπει επίσης να ληφθούν υπόψη όλοι αυτοί οι παράγοντες ε, κατά τη χάραξη και υιοθέτηση πολιτικών και στρατηγικών που στόχο έχουν την προστασία της οικονομίας. Ο αρνητικός αντίκτυπος των κλιματικών αλλαγών στις καλλιέργειες, ε, στην κτηνοτροφία και στην αλία λόγω της μεταβλητικότητας των μετεωρολογικών παραγόντων και συνθηκών υγρασία, θερμοκρασία, ακραία και καιρικά φαινόμενα όπως πλημμύρες, καύσονες, τύφωνας, ε, επίπεδο άλατος, οξύνηση, ξηρασίες και όλα αυτά θα πρέπει να ληφθούν υπόψη. Να σας δώσω ένα παράδειγμα από το Παγκλαντές. Οι πλημμύρες είναι μεγάλο πρόβλημα και έχουν οδηγήσει σε καταστροφή. Το 1998 είχαμε τεράστιες πλημμύρες στο 60% της χώρας με 1,2 δισεκατομμύρια ζημιές και 45 εκατομμύρια άστεγοι ως θύματα αυτών των πλημμυρών. Αυτό δείχνει μελέτη του Υπουργείου Περιβάλλοντος του Μπαγκλαντές το 2009. Επίσης, ε, ε, το 2018 ήταν το Μπαγκλαντές από τις ε, πιο τις χώρες που έχουν πληγεί περισσότερο από τα καιρικά φαινόμενα την τελευταία 20 ετία και η διάβρωση αφήνει εκατομμύρια συνανθρώπους μας άστεγους. Οπότε το κλίμα επηρεάζει αρνητικά το ΑΕΠ. Το Μπαγκλαντές ήδη έχει ένα σχέδιο για, ε, για την πολιτική μας μέχρι το 2100 και θα εφαρμόσουμε επενδυτικά προγράμματα που θα οδηγήσουν σε κοινωνική ανάπτυξη και σε αύξηση κατά 8% του ΑΕΠ αλλά θα πρέπει να λάβουμε υπόψη όλες τις ε, κλιματικές αλλαγές και το σχετικό προβληματισμό. Γιατί πολύ συχνά η επίθεση των μετεωρολογικών φαινομένων ε, έχει ως συνέπεια την αύξηση της φτώχειας και σίγουρα οι θεομηνίες ε, επηρεάζουν τους φυσικούς σπόρους και αυξάνουν τις οικονομικές ζημίες. Γι' αυτό και είναι επιτακτική ανάγκη η ανέβρεση κατάλληλου μηχανισμού για την καλύτερη προσαρμογή στις κλιματικές αλλαγές και τη χρηματοδότηση αυτής της προσαρμογής. Η χρηματοδότηση και η διαχείριση των πόρων θα είναι απαραίτητη παράγοντε για την ανέβρεση μια λύση στο πρόβλημα. Και θα σα παρουσιάσω κάποια μοντέλα που χρησιμοποιήσαμε στο Μπαγκλαντέ και τα εφαρμόσαμε. Το Μπαγκλαντέ έχει οθετήσει ε, ε, πολλά μέτρα για να συμπεριλάβουμε τις κλιματικές ε, αλλαγές στο πενταετές μας σχέδιο. Μια ολοκληρωμένη στρατηγική και σχέδιο δράση υπάρχει στον Μπαγκλαντέ. Επίση, εθνικά προγράμματα δράση και προσαρμογή στι κλιματικέ αλλαγέ. Έχουμε και ένα καταπιστευματικό ταμείο που συστήσαμε με ίδιου πόρου. Και μάλιστα αυτό έχει αναγνωριστεί από τον Πρωθυπουργό μα Γι' αυτό και έχει λάβει το βραβείο του ΟΗΕ πρωτοθλητής ε, της γης για το περιβάλλον. Επίσης, οι εθνικά καθορισμένες μας συνεισφορές ε, είναι πολύ υψηλές και το Μπαγκλαντές επηρέασε τις εθνικά καθορισμένες προσφορές μας ε, που είναι στοιχείο της Συμφωνίας του Παρισιού, παρόλο που είναι από τις πιο ευάλωτες χώρες και για μας η προσαρμογή είναι προτεραιότητα. Επίσης, έχουμε δεσμευθεί να κάνουμε τη μετάβαση στην οικονομία μας για να ε, μειώσουμε τις εκπομπές άνθρακα. Επίση, θα πρέπει να ενισχύσουμε τη χρηματοδότηση για να είμαστε ανθεκτικοί στι αλλαγέ του κλίματο. Κάτι που προποθέτει μια διαχείριση σε φορολογικό επίπεδο. Γιατί θα πρέπει να έχουμε μια σωστή δημοσιονομική διαχείριση που θα λαμβάνει υπόψη και τι κλιματικέ αλλαγέ. Θα πρέπει να ενισχυθεί η οικονομική διακυβέρνηση και να, συντονίσουμε την οικονομική μα διακυβέρνηση με άλλου φορεί που είναι αρμόδιοι για το περιβάλλον. Αυτά ήταν συντομία κάποια μέτρα που εθέτησε η κυβέρνηση του Μπαγκλαντέ και πολύ ευχαρίστω τα μοντέλα μας να σας τα παρουσιάσουμε αν υπάρχει ενδιαφέρον για περισσότερες λεπτομέρειες και το πώς λειτουργούν όλα αυτά τα μοντέλα. Πιστεύω ότι όλοι έχουμε πολλά να διδαχθούμε από τους συναδέλφους και μόνο έτσι θα δημιουργήσουμε αποτελεσματικές εταιρικές σχέσεις μεταξύ των κοινοβουλίων προκειμένου να αναπτύξουμε μια πραγματική κοινοβουλευτική περιβαλλοντική διπλωματία και να οδηγηθούμε σε μια παγκόσμια οικονομία που θα είναι ανθεκτική στις κλιματικές αλλαγές. Ευχαριστώ. Thank you. Ευχαριστώ όλους τους ομιλητές. Τώρα είναι η δική σας ευκαιρία να θέσετε ερωτήσεις ή να κάνετε κάποιο σχόλιο, αν θέλετε. Απλώς να πω ότι μόνο τα μέλη των κοινοβουλίων καλούνται να πάρουν το λόγο. Επομένως, η διαδικασία που θα ακολουθήσουμε είναι catch Όταν ε, κάποιος θέλει το λόγο, σε οποιοδήποτε στάδιο, παρακαλώ να σηκώσετε το χέρι σας, θα σας δώσουμε το λόγο. Και θα ήθελα να προτείνω να ξεκινήσετε με το να συστηθείτε πριν ε, αρχίσετε την παρέμβασή σας. Και μάλιστα ξέχασα και εγώ να συστηθώ στην αρχή. Λέγομαι Νίνα Αγγίλ και είμαι μέλος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου από τα Δυτικά Μίτλαντ στο Ηνωμένο Βασίλειο. Και επίσης είμαι και αντιπρόεδρος ε, της Αντιπροσωπείας για την Ινδία και επίσης είμαι και μέλος στην Αντιπροσωπεία για την Εσία και έχω συμμετέχει και στην ε, Επιτροπή ε, για την Κίνα. Μόλις επέστρεψα από την Κίνα και έχω εργαστεί πολύ και για το θέμα της Ινδίας. Να καλέσω τώρα τον κύριο Ράτσα να πάρει το λόγο που το ζήτησε πρώτος και στη συνέχεια ο κύριος που βρίσκεται ακριβώ πίσω του. Παρακαλώ. Αξιότιμη Πρόεδρε, αγαπητοί προσκεκλημένοι και μέλη του Κοινοβουλίου. για το θέμα του κλίματος και της οικονομίας. Βλέπουμε ότι η κλιματική αλλαγή πλήττει την παραγωγή, την υγεία και την οικονομία μας, όχι μόνο στην Ινδία, αλλά και σε άλλες χώρες. Αναφερθήκατε σε προβλήματα και εκτιμάμε ότι μπορούμε να έχουμε τεράστιες απώλειες. Φυσικά, μπορεί αυτό να αποδοθεί μόνο στην κλιματική αλλαγή. Και πάλι όμως, ένα μεγάλο ποσοστό του πληθυσμού στην Ινδία εξαρτάται από τη γεωργία και Μερικές φορές ε, έχουμε και πλημμύρες που καταστρέφουν τις καλλιέργειες. Και έχουμε πάρα πολλές συνεπίσεις όχι μόνο στον οικονομικό τομέα, αλλά και στην υγεία. Έχουμε πάρα πολλούς ανθρώπους που παθαίνουν καρκίνο και έχουμε και ψάρια σε λίμνες και σε ποτάμια που δηλητηριάζονται. Τα βρίσκουμε δηλητηριασμένα λόγω των λιμάτων. Και έχουμε ε, μια μεγάλη κρίση στο θέμα της διαχείρισης των αποβλήτων. Αυτό το θέμα είναι πολύ μεγάλο, τη διαχείριση των αποβλήτων και ο Πρωθυπουργό μας ανέλαβε μια πρωτοβουλία για να υπάρξει συμφωνία για το κλίμα. Και από τότε έχει μια παγιωμένη θέση. Υπάρχει μια αύξηση των προσπαθειών μας Αν δεν έχουμε βέβαια τη βοήθεια των αναπτυγμένων χωρών, δεν είναι εύκολο οι αναπτυσσόμενες χώρες να αντιμετωπίσουν τα κλιματικά ζητήματα. Το θέμα της μείωσης του άνθρακα. Πρέπει να έχουμε καθαρή τεχνολογία, χρηματοδότηση οικοδόμηση ικανοτήτων, και αν δεν υπάρξει υποστήριξη από εσά δεν είναι δυνατόν να τα καταφέρουμε. Μέχρι το 2022 έχουμε θέσει κάποιους στόχους Έχουμε και μία ατζέντα, μία στρατηγική δράσης. Βέβαια αυτά δεν έχουν προχωρήσει και ιδιαίτερα. Αυτή είναι η εκκλησία μου λοιπόν, μέσω της Ευρωπαϊκής Ένωσης έχετε μεγάλη επιρροή και πρέπει να την ασκήσετε γιατί τη χρειάζονται οι αναπτυσσόμενες χώρες. Η μείωση των εκπομπών έχει ψηφιστεί από το 2005 στο 2010 είχαμε 10% μείωση στις εκπομπές και η κυβέρνηση έχει θέσει ένα συγκεκριμένο στόχο για την καταπολέμηση της κλιματικής αλλαγής και τώρα θα έχουμε μια κρόαση Ουσιαστικά κάνουμε και μια μετάβαση προς μια ενέργεια που να μην προέρχεται από ρηκτά καύσιμα. Μέχρι το 2022 ο στόχος μας είναι να έχουμε ενέργεια 125 GB και σιγά σιγά θα εξαλείψουμε την ενέργεια από τα ορυκτά καύσιμα. Έτσι λοιπόν, κινούμαστε προς την καθαρή ενέργεια που δεν θα έχει επιπτώσει στο κλίμα. Βέβαια αυτό θίγει και την παραγωγή των τροφίμων σε πάρα πολλά μέρη της χώρας Μερικές φορές οι καλλιέργειες αντιστρέφονται ολοκληρωτικά. Αυτό δεν συνέβαινε στο παρελθόν. Όμως τα τελευταία χρόνια βλέπουμε να συμβαίνει αυτό το φαινόμενο πολύ συχνά και φυσικά θα πρέπει να το δούμε και αυτό το ζήτημα στα πλαίσια των πολυμερών συζητήσεων. Και οι ευρωπαϊκές χώρες πρέπει να ενθαρρύνουν τις συμπράξεις στον τομέα αυτό. βλέπουμε τώρα ότι υπάρχει συνειδητοποίηση ακόμη και σε επίπεδο grassroots, σε επίπεδο πολιτών. Επίσης αυτό βοηθά την οικονομική μετάβαση, την οικονομική μεταρρύθμιση. Εμείς ε, θέλουμε να καταπολεμήσουμε και την ε, φτώχεια και την ε, ανεργία που συνδέονται και με την κλιματική αλλαγή. Σας ευχαριστώ που μου δώσατε την ευκαιρία να αναφέρω τις απόψεις μου. Ευχαριστώ πολύ. Uh, Ευχαριστούμε πάρα πολύ για την παρέμβασή σας αυτή. Νομίζω ότι ένα από τα σχόλια τα οποία κάνατε και τα κρατάω είναι ότι χρειάζεστε υποστήριξη. Πρέπει λοιπόν να καθορίσουμε τι είδου θα είναι η υποστήριξη που θα παρασχεθεί προ τι αναπτυσσόμενε χώρε για να μειώσουν τι εκπομπέ. Ε, δεν ξέρω αν ίσως κάποιος από το πάνελ θα ήθελε να κάνει κάποιο σχόλιο για μεταφορά τεχνολογικής γνώσης για παράδειγμα τι πρέπει να παρασχεθεί στις αναπτυσσόμενες χώρες Πείτε μας σας παρακαλώ από το πάνελ αν θέλετε να τοποθετηθείτε. Δεν είναι ανάγκη αν δεν θέλετε, αλλά αν θέλετε βεβαίως μπορείτε να παρέμβετε στη συζήτηση. Βλέπω ότι η συνάδελφος από τις Φιλιππίνες ε, μου ζητά το λόγο. Παρακαλώ. Ευχαριστώ. Το... Η σύμβαση πλαίσιο του ΟΗΕ για την κλιματική αλλαγή ξεκαθαρίζει ε, τα ζητήματα γύρω από την τεχνολογία και την κλιματική αλλαγή και υπάρχει δίσμευση ε, δέσμευση οι αναπτυγμένες χώρες να παράσχουν στις αναπτυσσόμενες χώρες την τεχνολογία και τις γνώσεις, την εμπειρογνωμοσύνη για να μπορέσουν αυτές να υλοποιήσουν τις αναγκαίες προσαρμογές. Αυτό είναι σαφές. Ένα από τα αιτήματα που έχουμε λοιπόν και που διεκδικούμε είναι όλες οι άλλες παγκόσμιες συμφωνίες και συμβάσεις να αναθεωρηθούν ώστε να ενταχθεί και αυτή η απέτηση που προκύπτει από αυτήν την συμφωνία πλαίσιο. Για παράδειγμα, ένα τομέα στον οποίο πρέπει να υπάρξει επανεξέταση είναι οι εμπορικές συμφωνίες που έχουν συνευθεί σε διεθνές επίπεδο, διότι πολλές φορές αυτές εμποδίζουν την μεταφορά τεχνολογίας που ε, πλέον ε, έχει κατοχυρωθεί στην Σύμβαση για το Κλίμα. Είναι μία από τις δεσμεύσεις τις οποίες ε, έχουν αναλάβει τα συμβαλόμενα μέρη της Σύμβασης. Κυρία Τσάουντουρη από τον Μπαγκλαντές. Ευχαριστώ. Νομίζω ότι είναι πολύ σημαντική η διάσταση αυτή, διότι η χρηματοδότηση της ε, αντιμετώπισης κλιματικής αλλαγής ε, είναι ένα από τα πολύ σημαντικά εργαλεία που έχουμε στα χέρια μας προκειμένου οι, αναπτυγμένες, ε, οι αναπτυσσόμενες και οι λιγότερα αναπτυγμένες χώρες να ανταποκριθούν στην, στις υποχρεώσεις τους. Στο πλαίσιο λοιπόν της συμφωνίας πλαίσιο του Ταμείου για την Πράσινη Ανάπτυξη, τη συμφωνία των Παρισίων. Ε, υπάρχουν τέτοιες διατάξεις, ε, όμως αυτή τη στιγμή δεν υπάρχει επαρκής χρηματοδότηση. Πρέπει να δοθούν περισσότερα κίνητρα ε, οι αναπτυσσόμενες χώρες να χρηματοδοτήσουν, οι ανεπτυγμένες χώρες μάλλον να βοηθήσουν τις αναπτυσσόμενες χώρες να ανταποκριθούν στις υποχρεώσεις τους. Μήπως λοιπόν το, η σημερινή μας διάσκεψη είναι ένα καλό εργαλείο ώστε να παρακινηθούν εκείνοι που έχουν αναλάβει αυτές τις δεσμεύσεις στις υποχρεώσεις τους να προχωρήσουν ε, δηλαδή σε, σε όσα είναι αναγκαία να κάνουν. Να πω ότι ε, είναι θετικό το γεγονός ότι αναφερθήκατε στο Ταμείο για το Πράσινο Κλίμα γιατί εγώ ε, είμαι παρατηρήτρια και συμμετέχω στο Διοικητικό Συμβούλιο εκ μέρους των μη κυβερνητικών οργανώσεων. Ε, πρέπει να σας πω λοιπόν ότι τα χρήματα που έχουμε στο προπολογισμό μας τελειώνουν και γι' αυτό μία από τις εκκλήσεις μας είναι ε, οι ανεπτυγμένες χώρες να συνεισφέρουν στον προϋπολογισμό του πράσινου αυτού ταμείου και αυτό πρέπει να γίνει το συντομότερο δυνατό. Ευχαριστώ. Ο συνάδελφος από το Πακιστάν έχει το λόγο. Γεια σας, Σεβελ Τζάβεντ, βουλευτής από το Πακιστάν και μέλος της Μόνιμης Επιτροπής για την Κλιματική Αλλαγή. Χαίρομαι πολύ που συμμετέχω σε αυτήν την κοινοβουλευτική συνδιάσκεψη Ευρώπης-Ασίας που ε, θεωρώ ότι αποτελεί ένα μήνυμα ότι μέσω της συνεργασίας μας μπορούμε να αντιμετωπίσουμε την κλιματική αλλαγή, να κάνουμε τον κόσμο μας καλύτερο για τις μελλοντικέ γενιές. Το Πακιστάν έχει κάνει μεγάλες θυσίες για την παγκόσμια ειρήνη, για το παγκόσμιο περιβάλλον και βεβαίως για το περιβάλλον σε συνδυασμό με την ειρήνη. Οι μεγάλοι ηγέτες, όπως λέγεται, δεν έχουν το βλέμμα του στραμμένο στις εκλογές, αλλά στις επόμενες, τις μελλοντικέ γενιές. Και εδώ ένα παράδειγμα από το Πακιστάν, υπό την ηγεσία του Ιμραν Καν, το Πακιστάν είναι η πρώτη χώρα που ε, ανταποκρίθηκε ε, στην ε, διεθνή της δέσμευση για αναδάσωση Έχουμε ε, φυτέψει πάνω από ένα δισεκατομμύριο δέντρα, κάτι που βοήθησε το Πακιστάν να προσελκύσει ιδιωτικές επενδύσεις και ε, ενίσχυσε τα τοπικά εισοδήματα, δημιούργησε πάνω από 500.000 θέσεις ε, εργασίας στον οικολογικό τομέα. Και αυτό με την, με την στήριξη του IUCN που μας ε, παρήχε 150 ε, εκατομμύρια εκτάρια έως το 2020 και 350 έως το 2030. Το Πακιστάν λοιπόν είναι η πρώτη χώρα που ανταποκρίθηκε στην υποχρέωσή της να αναδασώσει ε, τεράστιες εκτάσεις. Και με τον έλεγχο του WWF αποδείχθηκε ότι το project αυτό είχε σημαντικότατη κοινωνική, οικονομική και περιβαλλοντική επιτυχία. Το ίδιο αναγνώρισε και το Παγκόσμιο Οικονομικό Φόρουμ. Το επόμενο σχέδιο της κυβέρνησης του Πακιστάν είναι να φυτέψει πάνω από 10 δισεκατομμύρια δέντρα σε ολόκληρη την επικράτεια του Πακιστάν και την ημέρα έναρξης του προγράμματος αυτούς, αυτού ε, φυτέψαμε 1,5 ε, εκατομμύρια δέντρα. Ελπίζουμε λοιπόν τα επόμενα πέντε χρόνια να φυτέψουμε 10 δισεκατομμύρια δέντρα. Τα μέτρα πολιτικής μας εστιάζονται στις καθαρές μορφές ενέργειας, στις πράσινες θέσεις απασχόλησης και θεωρούμε ότι η απέτηση για 25% δασική κάλυψη, εμείς αυτή τη στιγμή ε, έχουμε καλύψει μόλις το 2,5% αυτού του στόχου. Γι' αυτό και επικεντρωνόμαστε σε αυτό, να υπάρξει μια μεταστροφή στην οικονομία, καθαρή ενέργεια, καθαρό νερό, πράσινες θέσεις εργασίας, αποτελεσματική χρήση των φυσικών μας πόρων. Μαζί θεωρούμε ότι μπορούμε και πρέπει να καταπολεμήσουμε την κλιματική αλλαγή. Και από αυτό το βήμα εμείς πρέπει να σας πω ότι αντλούμε πολλά διδάγματα, ακούμε πολύ σημαντικές και ενδιαφέρουσες ιδέες και βλέπω ότι υπάρχει μεγάλη σοβαρότητα ως προς ε, το πώς αντιμετωπίζουμε τις προκλήσεις αυτές. Σας εύχομαι λοιπόν κάθε επιτυχία, σας ευχαριστώ πάρα πολύ που μας προσκαλέσατε, σας ευχαριστούμε πολύ που μας ακούτε γιατί θεωρώ ότι κομίζουμε ένα μήνυμα για το πώς η πολιτική βούληση μπορεί να συμβάλλει στην επίτευξη σημαντικότατων ε, οροσίμων και ένα από αυτά τα ορόσημα είναι αυτό που σας μετέφερα εδώ για τη φύτευση 10 δισεκατομμυρίων δέντρων στο Πακιστάν. Ευχαριστούμε πολύ για τη δήλωση αυτή. Μας ενθαρρύνετε με αυτά που λέτε, πρέπει να σας πω. Περνάμε τώρα στον εκπρόσωπο του Λάος. Αξιότιμη συμπρόεδρε, ονομάζομαι Κιν Τόγκ Σινκ, μέλος του Εθνικού Κοινοβουλίου του ΛΑΟΣ. Εκ μέρους της αντιπροσωπείας μας θα ήθελα να εκφράσω τις ειλικρινείς ευχαριστίες μου για τη διοργάνωση αυτής της δέκατης Ευρωασιατικής Κοινοβουλευτικής Συνέλευσης και να σας συγχαρώ για την άρτια διοργάνωση. Θα θέλαμε και εμείς ε, να σας ευχαριστήσουμε επίσης για τη θερμή υποδοχή και φιλοξενία που επιφυλάξατε στην αντιπροσωπεία μας. Κυρία Πρόεδρε, είναι πολύ σημαντικό το αντικείμενο της σημερινής συζήτησης. Οι κλιματικές αλλαγές, το περιβάλλον και ο αντίκτυπό του στην οικονομία ε, είναι θέμα που απασχόλησε πολλές ε, περιφερειακές ε, και διεθνείς διασκέψεις τα τελευταία χρόνια και έχουν γίνει πολύ επίκαιρο ζήτημα. Τα αποτελέσματα του αντίκτυπου των κλιματικών αλλαγών είναι ορατά σε κάθε γωνιά του πλανήτη, ακόμη και στη δική μου πατρίδα, το Λάος. Οι κλιματικές αλλαγές είναι από τις πρωταρχικές προκλήσεις των καιρών μας και μία από τις σημαντικότερες προκλήσεις της κοινωνίας μας είναι το περιβάλλον, η προστασία του περιβάλλοντος. Και μάλιστα οι συνέπειες των κλιματικών αλλαγών ε, συνιστούν απειλή και για την παραγωγή τροφίμων, ε, γιατί ε, η αύξηση του επίπεδου της θάλασσας έχει οδηγήσει σε καταστροφικές πλημμύρες. οι κλιματικές αλλαγές είναι πραγματικότητα. Και θα ήθελα θα σας, να σας αναφέρω ένα παράδειγμα από το Λάος. Οι τροπικές καταιγίδε που ξεκίνησαν λόγω των χαμηλών πιέσεων σε μια θάλασσα πολύ μακριά από το Λάος προκάλεσαν σοβαρότατες πλημμύρες και μάλιστα και οι 18 επαρχές του Λάος έχουν πληγεί από τις πλημμύρες αυτές, έχουν υποστεί σοβαρές ζημίες, πολλό δε μάλλον που συνεχίζονται ισχυρές βροχοπτώσεις. Λόγω των κατολιστήσεων και των πλημμυρών σε 16 ε, επαρχίες αλλά και στην πρωτεύουσα είχαμε τρομερές ζημίες 100 πόλεις, 299 χωριά και ε, χιλιάδες οικογένειες έμειναν άστεγες και 54 άτομα έχασαν τη ζωή τους ενώ εκατοντάδες ε, είναι οι αγνοούμενοι αυτών των πλημμυρών. 20.500 άνθρωποι χρειάστηκαν να εκτοπιστούν εσωτερικά και αυτές ήταν και μάλιστα οι σοβαρότερες πλημμύρες οφείλονται στην κατάρρευση ενός φράγματος ε, ενός υδροηλεκτρικού σταθμού κοντά στο Νόη. Στις 31 Ιουλίου του 2018, κάτι που προκάλεσε το θάνατο 40 συνανθρώπων μας και 97 ε, αγνοούνται, ενώ 6.600 χρειάστηκε να ε, εκτοπιστούν εσωτερικά. Και σίγουρα ε, η μικρή οικονομία του Λάος ε, λόγω αυτών των πλημμυρών έχει υποστεί μεγάλες ζημίες. Το ίδιο και ο κοινωνικός ιστός. 9.345 οικογένειες χρειάστηκε να στεγαστούν λόγω της ζημίας που υπέστησαν οι δικές τους κατοικίες. Μάλιστα επηρεάστηκαν ε, και υπηρεσίες ε, υγείας και εκπαίδευσης. 4.600 σταθμοί καθαρισμού, βιολογικού καθαρισμού έχουν πληγεί. 8.000 μέτρα αποχευτικού συστήματος και πολλές χιλιάδες σχολεία καταστράφηκαν. 460 δρόμοι και 52 γέφυρες ε, έχουν καταστραφεί ή παρασυρθεί από τα ύδατα των πλημμυρών. Στη Γεωργία περίπου 114.000 ε, εκτάρια οριζόνων, 3.400 σταθμοί δατοκαλλιέργειας και 2.000 ε, βοηδοί και 1.000 χείρι και 30.000 ε, πουλερικά θανατώθηκαν από τις πλημμύρες. Εξαιτία αυτών των σοβαρότητων ζημιών που είχαμε και στο ε, δίκτυο ηλεκτροδότησης, οι απώλειες ήταν πολλές. Οπότε είναι εμφανές ότι οι κλιματικές αλλαγές είναι παγκόσμιο ζήτημα και επηρεάζει κυρίως ε, αρνητικά και πλήττει τους πιο ευάλωτους συνανθρώπους μας στις πιο φτωχές χώρες. Γι' αυτό θα ήθελα να εκφράσω με την ευκαιρία αυτή τις βαθύτερες ευχαριστίες μας και την ευγνωμοσύνη μας προς όλες τις χώρες, τους αναπτυξιακούς μας εταίρους και τις διεθνείς οργανώσεις για τη συμπαράσταση και την ανθρωπιστική αρρωγή που παρήχαν στο λαό του Λάος και κυρίως σε όσους ε, επηρεάστηκαν από την κατάρρευση του φράγματος στον υδροηλεκτρικό σταθμό κοντά στο Νόη. Το λαός αποδίδει ιδιαίτερη σημασία στο θέμα των κλιματικών αλλαγών. Έχουμε θετήσει μάλιστα μία φιλοπεριβαλλοντική πολιτική και μέχρι το 2020 το 70% της επικράτησης του ΛΑΟΣ θέλουμε να καλύπτεται από δάση. Και το Μάιο του 2015 εκδώσαμε ένα διάταγμα που απαγορεύει την εξαγωγή ξύλου και την εξαγωγή της προϊόντων υλοτομίας. Έχουμε κινητοποιηθεί ε, σε όλη μας την επικράτεια και μάλιστα έχουμε ε, κυρώσει πολλές διεθνείς συμβάσεις για τις κλιματικές αλλαγές όπως τη Διεθνή Σύμβαση για τις κλιματικές αλλαγές του 1995, το πρωτόκολλο του Κιώτο το 2003 και τη Συμφωνία των Παρισίων. Μάλιστα έχουμε και το εθνικό σχέδιο προσαρμογής και δράσης για τις κλιματικές αλλαγές. Και έχουμε και ένα νόμο για τη διαχείριση των θεομηνιών και τις κλιματικές αλλαγές που, που απορρέει από κάποιες διεθνείς συμβάσεις. Και αυτό θα είναι καλό σημείο αναφοράς για, τη, για το νομοθετικό μας πλαίσιο και την διεθνή μας συνεργασία στο μέλλον. Το Λάος ήταν ανέκαθεν υπέρ του ενεργού ρόλου της ΑΣΕΠ και των ευρασιατικών χωρών και θεωρούμε ότι μπορούμε να ενισχύσουμε την πολυμερή συνεργασία. Και γι' αυτό η Εθνική μας Συνέλευση θα διοργανώσει την επόμενη διάσκεψη στη χώρα μας. Θα θέλαμε να διατρανώσουμε την προσήλωσή μας στα ζητήματα των κλιματικών αλλαγών και του περιβάλλοντος και απότερος μας στόχος είναι να δημιουργήσουμε τις απαραίτητες προϋποθέσεις ώστε να διαφυλάξουμε το περιβάλλον και να προωθήσουμε την ευρωασιατική εταιρική σχέση στα ζητήματα του περιβάλλοντος, προωθώντας τις διαπροσωπικές σχέσεις για να ζήσουμε όλοι ειρηνικά και να προωθήσουμε μια βιώσιμη οικονομική ανάπτυξη, ε, απασχόληση και αυξανόμενο βιωτικό επίπεδο για όλους. Ευχαριστώ. Uh, uh, uh, my η σειρά μου να συντονίσω τους επόμενους τρεις ομιλητές. Επειδή περνάει ο χρόνος, ας περάσουμε στον επόμενο ομιλητή από την Ορβηγία. It has been really interesting to be here and listen to... Ήταν ε, πάρα πολύ ενδιαφέρον ε, που σας άκουσα όλους. Είδαμε ότι η Ασία και η Ευρώπη έχουν πολλές από τις ίδιες προκλήσεις. Σας παρακαλώ να παρουσιαστείτε. Προέρχομαι από το Νορβηγικό Κοινοβούλιο, από το κόμμα ε, της Πρόοδου όταν ε, αντιμετωπίσουμε το θέμα της κλιματικής αλλαγής και της οικονομίας ε, θα πρέπει να τονίσω καταρχήν τη σημασία του να διαφυλάτουμε τους κανόνες του πολυμερού συστήματος εμπορίου του ΠΟΕ. Δεν υπάρχει κανένα άλλο τρόπο να διασφαλίσουμε ότι οι αρχέ τη βιωσιμότητα του ανοιχτού και ανοιχτού εμπορίου εφαρμόζονται ομοιόμορφα στο διεθνέ εμπόριο. Αυξανόμενο προστατευτισμό και αυτό που φαίνεται να είναι ένα αναδυόμενο εμπορικό πόλεμο μπορεί να έχει ένα πολύ αρνητικό αντίκτυπο στην παγκόσμια οικονομία. Τέτοιε προοπτικέ είναι σοβαρέ, ιδίω όταν χρειάζεται να δημιουργήσουμε περισσότερε θέσει εργασία, να προσαρμόσουμε τα επιζήμια αποτελέσματα τη κλιματική αλλαγή και να διασφαλίσουμε τη βιωσιμότητα και την ε, ανάπτυξη όπου συμμετέχουν όλοι. Επιτρέψτε μου να ευστήσω την προσοχή σας σε μια πρωτοβουλία που ξεκίνησε στον Ταβός νωρίτερα φέτος από την Πρωθυπουργό της Νορβηγίας, Έρνα Σόλβερκ συμμετείχε σε ένα πάνελ υψηλού επίπεδου, ε, μάλλον δημιούργησε ένα πάνελ υψηλού επίπεδου για την οικοδόμηση μια βιώσιμη οικονομία των ωκεανών και συναντήθηκε το πάνελ για πρώτη φορά κατά τη διάρκεια τη 73η συνέλευση του ΟΗΕ την Δευτέρα αυτή την εβδομάδα. Ο παγκόσμιος πληθυσμός θα αυξηθεί το 2050 και ε, για να καλύψουμε τις ανάγκες ε, του πληθυσμού περισσότερο από τα τρόφιμά μας ενέργεια, φάρμακα, ορυκτά και μεταφορές θα πρέπει να έρχονται από τους ωκεανούς. Έτσι λοιπόν χρειαζόμαστε μια βιώσιμη ανάπτυξη στις παγκόσμιες βιομηχανίες των ωκεανών ε, για να στους κλάδους του ωκεανού δημιουργήσουμε θέσεις εργασίας, εισόδημα, οικονομική και κοινωνική ανάπτυξη. Επομένως είναι ε, ζωτικό ε, τα κράτη, ε, τα θαλάσσια στην Ευρώπη και στην Ασία να συνεργαστούν για να τονίσουν το τεράστιο δυναμικό που βρίσκεται στο να οικοδομήσουμε μια βιώσιμη οικονομία των ωκεανών. Αυτό σημαίνει να διασφαλίσουμε καθαρούς και υγιείς ωκεανούς βάσει της πρότασης της Νορβηγίας η συνέλευση περιβάλλοντος του ΙΕ έχει οθετήσει ένα όραμα για ε, μηδενικά πλαστικά απόβλητα στους ωκεανούς. Η Νερβηγία έχει ξεκινήσει ένα πρόγραμμα που στοχεύει στο να καταπολεμήσουμε τα μικροπλαστικά και τα ε, σκουπίδια στους ωκεανούς σε αναπτυσσόμενες χώρες, πολλά από τα οποία προέρχονται από τα ποτάμια. Ελπίζουμε ότι θα συνεργαστούμε με πολλές χώρες παγκοσμίω και με πολλές χώρες στην Ασία για να επιλύσουμε αυτή την πρόκληση. Thank you. very much for your... Ευχαριστώ πολύ για τη δήλωσή σας. Θα δώσω το λόγο στον επόμενο μιλητή από τη Φιλανδία, παρακαλώ. ένα μήνυμα για τους εταίρους μας ε, από την Ασία. Είχα μια ερώτηση βέβαια που απαντήθηκε εν μέρη, αλλά παρόλα αυτά να κάνω ένα σχόλιο. Ποια είναι η άποψή σας αν διάφουμε, δούμε διάφορα εργαλεία εναλλακτικέ για το πώς θα μειώσουμε τις εκπομπές διοξιδίου του άνθρακα στις χώρες σας. Αν έχουμε τρεις διαφορετικές επιλογές καταρχήν λύση που να βασίζεται στην αγορά. Η μία θα μπορούσε να είναι ένα σύστημα εκπορίας εκπομπών, όπως έχουμε στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Ένα δεύτερο θα μπορούσε να είναι η ρύθμιση. Νομοθετική ρύθμιση. Δηλαδή, στην νομοθεσία θα ορίζεται τι επιτρέπεται και τι όχι. Αυτή είναι μια άλλη εναλλακτική. Και τρίτη εναλλακτική στην ερώτησή μου είναι συνεργασία της τεχνολογίας συνεργασία με την τεχνολογία προκειμένου να μειωθούν οι εκπομπές διεξιδίου του άνθρακα. Ποιο από όλα αυτά θεωρείτε ως πιο ελκυστικό τρόπο για να προχωρήσετε στις ε, ασιατικές χώρες. Και θα ήθελα να στρεφώ σε κάποιους από τους ε, Ασιάτες εταίρους που βρίσκεται στο βήμα. Για να μου απαντήσετε. Πιστεύω ότι η εμπειρία της εφαρμογής του πρωτοκόλλου του Κιώτο μας δείχνουν ότι οι προσεγγίσεις ε, που έχουν να κάνουν με, που βασίζονται στην αγορά δεν είναι αποτελεσματικές και αυτή είναι μια πολύ έντονη συζήτηση σε διεθνές επίπεδο γιατί υπάρχουν ε, πολλές προσεγγίσεις που δεν βασίζονται στην αγορά και είναι επιτάπητος και γίνεται, δίνεται μεγάλη μάχη για το αν θα πρέπει να υπάρχει επέκταση των προσεγγίσεων που βασίζονται στην αγορά ή αν θα πρέπει να έχουμε μία αποφασιστική προσαρμογή των προσεγγίσεων που δεν βασίζονται στην αγορά. Για μας το πιο αποτελεσματικό θα ήταν ε, η μέθοδη να μετατραπούν τα συστήματα ενέργειας από τα ορυκτά καύσιμα στις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Και δεν νομίζω ότι δεν είναι το ένα ή το άλλο. Χρειαζόμαστε νομοθεσία που θα δώσει στις κυβερνήσεις την όθηση αυτή, δηλαδή να αναγκαστούν οι κυβερνήσεις, κυρίως το εκτελεστικό, να αναλάβει όλα τα απαραίτητα μέτρα και να κάνει τα απαραίτητα βήματα προκειμένου να έχουμε αυτή την ενεργειακή μετάβαση. Και γι' αυτό χρειαζόμαστε νομοθεσία έτσι ώστε να είμαστε σίγουροι ότι θα υπάρχουν ε, ανώτατα όρια, ότι θα υπάρχουν ε, υπεραίτητοι πόροι και θα υπάρχει και απαραίτητο χρονοδιάγραμμα για την εξάλληψη. Και επίση ε, η νομοθεσία θα μπορούσε να καταρτήσει ένα χρονοδιάγραμμα για να σταματήσει η περαιτέρω επέκταση τη χρήση ορυκτών καυσίμων. Γιατί ξέρετε, σε κάποιες χώρες στην Ασία μπορεί να υπάρχουν ε, φιλοδοξίες για να πετύχουν τους στόχους ε, των Παρισίων. Πολλές ε, χώρες βασίζονται και επεκτείνουν τα σχέδιά τους για ενέργεια ρηκτά καύσιμα. Έχουμε εκατοντάδες τέτοια εργοστάσια σε όλη την Ασία. Έτσι λοιπόν πρέπει να έχουμε σαφή νομοθεσία για να δυσφαλίσουμε ότι υπάρχει πολιτική βούληση. Το δεύτερο είναι η τεχνολογική συνεργασία και αυτό βέβαια είναι πολύ σημαντικό. Νομίζω ότι έχει γίνει σημαντική πρόοδος από την Κίνα, παραδείγματο χάρη, στην ε, ε μεγέθυνση της, ε, του κλάδου της ηλιακής ενέργειας και θα πρέπει να υπάρχει τεχνολογική συνεργασία γιατί οι άλλες συμφωνίες, κυρίως υπό τον Παγκόσμιο Οργανισμό Εμπορίου, είναι συμφωνίες που αποτελούν εμπόδια Γι' αυτό και η κινέζικη εμπειρία είναι ένα παράδειγμα. Επομένως, θα πρέπει να υπάρχει σαφής πολιτική βούληση για να μην υπάρχουν εμπόδια για την ε, τεχνολογική μετάβαση και για τη χρήση και την εφαρμογή τεχνολογιών που θα επιτρέψουν κάτι τέτοιο. Γι' αυτό τα δικαιώματα πνευματικής διοκτησίας ή ε, διεθνείς συμφωνίες για τα δικαιώματα ε, πνευματικής διοκτησίας για διπλώματα ευρεσιτεχνίας θα πρέπει να αναθεωρηθούν. Uh, Ευχαριστούμε. Είναι πολύ ενδιαφέρον το ερώτημα που θέτετε. Και μιας και ζητήσατε απάντηση από ασιατική σκοπιά, με χαρά μου να σας πω ότι συμφωνώ με την εμπειρογνώμονα. Δεν νομίζω ότι το ερώτημα πρέπει να τίθεται διαζευκτικά. Πρέπει να ε, συνδυάσουμε όλες τις πιθανές και δυνατές προσπάθειες για να δώσουμε απάντηση στις προκλήσεις. Αφενό λοιπόν ναι χρειάζεται νομοθετική ρύθμιση διότι χωρίς ρυθμιστικό και νομοθετικό πλαίσιο θα είναι πάρα πολύ δύσκολο να επιτύχουμε όλα όσα θέλουμε. Άρα είναι αναμφισβήτητο ότι το να έχει κανείς την κατάλληλη νομοθεσία είναι απαραίτητο. Υπάρχει επίσης ανάγκη να διευκολυνθούν οι μεταφορές τεχνολογίας, η οικοδόμηση ικανοτήτων, η χρηστή δημοσιονομική διαχείριση, η χρηματοδότηση, αλλά και η συμπερίληψη αυτών των στόχων στα εθνικά σχέδια ανάπτυξης. Όλα αυτά είναι εργαλεία που θα μπορούσαν να βοηθήσουν και ακόμη και αν ε, δεχόμαστε ότι δεν, υπάρχουν, δεν υπάρχει πανάκια είναι αναγκαίο να λαμβάνονται υπόψη βεβαίως όλες οι κοινωνικές, οικονομικές ε, περιστάσεις που επικρατούν σε κάθε χώρο. όλα αυτά, μέσω της συνεργασίας μπορούμε να προσδιορίσουμε τους ε, ζωτικής σημασίας τομείς, να εντοπίσουμε τις αιτίε των προβλημάτων και στη συνέχεια να διαμορφώσουμε τις λύσεις που θα χαρακτηρίσουν τις ε, κοινέ μας προσεγγίσεις για το τρόπο με τον οποίο θα επιλύσουμε τα προβλήματα και θα αντιμετωπίσουμε τις προκλήσεις μας για την περίπτωση της Κίνας θέλω να σας μιλήσω εγώ. Προσωπικά έχω την αίσθηση ότι συμφωνώ καταρχάς με τους εμπειρογνώμονες ότι η αγορά δεν είναι κατάλληλο εργαλείο. Κάτι που είναι πολύ ζωτική σημασίας για εμάς στην Κίνα είναι η πολιτική ηγεσία και το πολιτικό σύστημα. Ο σοσιαλισμός διαδραματίζει σημαντικότατο ρόλο. Ξέρετε ότι η Κίνα έχει ένα πολύ συγκεντρωτικό πολιτικό σύστημα. Και εγώ προσωπικά πιστεύω ότι αυτό αποτελεί σημαντικότατο παράγοντα για να εξασφαλίζεται η πρόοδος στους τομείς αυτούς. Θα ήθελα να σας ε, ρωτήσω κύριε Πρόεδρε. Είναι αλήθεια αυτά που αναφέρουν πολλά διεθνή μέσα μαζικής ενημέρωσης όπως το BBC ότι ε, δορυφορικές εικόνες αποδεικνύουν ότι αυτή τη στιγμή οικοδομούνται, κατασκευάζονται εκατοντάδες λιγνητορυχία σε ολόκληρη την επικράτεια της Κίνας. Μπορείτε να το επιβεβαιώσετε αυτό ως πληροφορία. Συγγνώμη, δεν κατάφερα να παρακολουθήσω το ερώτημά σας, λέει ο Πρόεδρος. Επαναλαμβάνω λοιπόν. Σε διεθνή μέσα μαζικής ενημέρωσης αναφέρεται η είδηση και παρατίθεται και δορυφορικές εικόνες οι οποίες δείχνουν ότι αυτή τη στιγμή στην Κίνα ε, κατασκευάζονται εκατοντάδες ε, ορυχεία ε, άνθρακα και εργοστάσια παραγωγής ηλεκτρισμού από άνθρακα. Εγώ προσωπικά ε, την συγκεκριμένη είδηση την παρακολούθησα στο BBC. Μπορείτε να το επιβεβαιώσετε. Πρόεδρος, δεν μπορώ να σας πω τίποτα γι' αυτό, γιατί δεν έχω καμία πληροφορία σχετική. Αν πράγματι ε, διαπιστωθεί ότι κάτι τέτοιο ισχύει, ε, σας διαβεβαιώ ότι θα λάβουμε μέτρα για να το αντιμετωπίσουμε. Αλλά αυτή τη στιγμή δυστυχώς δεν έχω κάποια σχετική ενημέρωση. Σας ευχαριστώ πάντως για το ερώτημα. Okay. All right, now let's move to the next. Ας περάσουμε τώρα στον επόμενο ομιλητή από την Ινδονησία. μπορεί να μιλήσει τη μητρική της γλώσσα γιατί υπάρχει διερμηνία. Σας ευχαριστώ. Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι. Honorable Chairperson. Αξιότιμοι συμπρόεδροι και μέλη της ΑΣΕΠ. parlemen Eropa untuk menjadi tuan rumah pertemuan kemitraan parlemen ASEAN Eropa ke-10. First of all, θα ήθελα πρώτα απ' όλα να εκφράσω τις ευχαριστίες μας προς, την, προς το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο για τη διοργάνωση της δέκατης αυτής ε, διακοινοβουλευτικής συνέλευσης ΑΣΕΠ. Of the Republic Indonesia Indonesia. Bahasa Inggris tadi. Εκπροσωπώ τη Δημοκρατία της Ινδονησίας. Diskusi hari ini, saya ingin menyampaikan beberapa poin pandangan. To contribute to today's... Θέλουμε και εμείς να συμβάλλουμε στη σημερινή συζήτηση με τα εξής σχόλια. Sebagai pandangan global bahwa perubahan iklim merupakan tantangan multimediasi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 Indonesia shares the... Και η Ινδονησία πιστεύει ότι οι κλιματικές αλλαγές είναι μια πολυδιάστατη πρόκληση και χρήζει πολυδιάστατης προσέγγισης στη χάραξη πολιτικής ε, για το μετριασμό των αρνητικών αποτελεσμάτων. Σε ό,τι αφορά την οικονομία, θεωρούμε ότι μπορούμε να συμφιλειώσουμε την οικονομική ανάπτυξη με την επιτεκτική ανάγκη της βιωσιμότητας του περιβάλλοντος. Η κυβέρνηση της Ινδονησίας ε, κάνει ό,τι μπορεί για να ευθυγραμμίσει τις εθνικές πολιτικές με τις παγκόσμιες προκλήσεις της πράσινης ανάπτυξης. Για παράδειγμα, έχουμε την Εθνική Πολιτική RTD+. Το 2015 ε, έχουμε πάγωμα των αδειών για τα δάση και τους τυρφώνες. Ε, έχουμε παρατείνει αυτό το δικαιοστάσιο προκειμένου να βελτιώσουμε την, το σχεδιασμό για τη χρήση γης και να ενισχύσουμε τα συστήματα πληροφορίας και συγκέντρωσης πληροφοριών δημιουργώντας ε, ε, φορείς και θεσμούς που θα μας επιτρέψουν να τηρήσουμε τους στόχους μας για μείωση των εκπομπών διοξιδίου του άνθρακα. Contoh lain adalah upaya kami untuk meningkatkan keberlanjutan minyak sawit kami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 tata kelola perkebunan kelapa sawit dan instrumen uji tuntas hak asasi manusia dalam industri minyak sawit di Indonesia. Another example. Ένα άλλο παράδειγμα των προσπαθειών μας να βελτιώσουμε τη βιωσιμότητα του φινικελαίου μας. Ε, εκτός ότι ενισχύσαμε τα, τις ε, αυστηρές προδιαγραφές για την παραγωγή φινικελαίου που συν, συνδέονται με τι διεθνεί προδιαγραφέ. Έχουμε και διορθωτικά μέτρα για το δικαιοστάσιο σε ό,τι αφορά την επέκταση τη γη για την καλλιέργεια αφήνικόδοντρων. Και μάλιστα έχουμε ε, προσπάθεια ανάκτησης των τριφώνων και ε, προσπάθεια για χρηστή βιώσιμη διαχείριση των φοινικοκαλλιεργειών και μάλιστα αυτή τη στιγμή εξετάζεται στη Βουλή μας ο σχετικός νόμος για τη φινικοκαλλιέργεια. Θέλουμε να ενισχύσουμε τη διακυβέρνηση στις φινικοκαλλιέργειες λαμβάνοντας υπόψη το σεβασμό των ανθρωπίνων δικαιωμάτων στον κλάδο της παραγωγής φινικελαίου. harapan terbaik kami untuk menyelamatkan lingkungan dan mengurangi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 terbaik menuju berkelanjutan energi keamanan diversi divers diversifikasi Renewable energy continues to be our... Οι ανανεώσιμες πηγές ενέργειας είναι ε, η ελπίδα μα για να σώσουμε το περιβάλλον και να μειώσουμε τι εκπομπέ εκπομπές διεξουδίου του άνθρακα τηρώντας του παγκόσμιου μα περιβαλλοντικού στόχου. Με φιλοπεριβαλλοντικέ στρατηγικέ για την ενέργεια θα συμβάλλουμε στην ανάπτυξη οικονομία και στη δημιουργία θέση απασχόληση. με βάση ε, την παγκόσμια ε, οργάνωση για τι ανανεώσιμε πηγέ ενέργεια 7,7 εκατομμύρια απασχολούνται στον κλάδο και στο Κοινοβούλιο της Ινδονησίας θεωρούμε ότι θα πρέπει να αναβαθμίσουμε τις προσπάθειές μας και να αυξήσουμε την συνειδητοποίηση της σημασίας που έχει ανανεώσιμη και βιώσιμη ενέργεια. Και μάλιστα πρόσφατα είχαμε το δεύτερο Παγκόσμιο Κοινοβουλευτικό Φόρουμ για τη βιώσιμη ανάπτυξη που ε, περιστρέφεται γύρω από το θέμα της εταιρική σχέσης για τη βιώσιμη ενέργεια για όλους. Και το φόρουμ αυτό αποτέλεσε πρωτοβουλία της Ινδονησίας και μάλιστα αυτή τη στιγμή είναι το μόνο παγκόσμιο διακοινοβουλευτικό φόρουμ για τους αναπτυξιακούς στόχους της χιλιετίας και ε, είχαμε κοινοβουλευτικούς από 46 χώρες που συζήτησαν και αντάλλαξαν τις βέλτιστες πρακτικές ό,τι αφορά την βιωσιμότητα της ενέργειας ε, και τη διαφοροποίηση των πηγών ενέργειας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 Tuhan untuk mempercepat negara EGA sehingga akan siap pada waktunya untuk mendukung kesepakatan Paris tentang uh, perubahan iklim dan tujuan pembangunan berkelanjutan. Trade plays a significant... Το εμπόριο διαδραματίζει σημαντικό ρόλο στην οικονομία και όπως όλες οι οικονομικές δραστηριότητες και το, και το εμπόριο σχετίζεται με τις εκπομπές αερίων του θερμοκηπίου. Θα πρέπει λοιπόν να έχουμε πρόσβαση σε φιλοπεριβαλλοντικέ τεχνολογίες, αγαθά και υπηρεσίε για να μπορέσουμε να κάνουμε τη μετάβαση προς μια οικονομία με χαμηλέ εκπομπές άνθρακα. Ένα μέτρο που υιοθετήσαμε είναι αύξηση του εμπορίου περιβαλλοντικών αγαθών και μάλιστα στα πλαίσια του ΠΟΕ γίνονται διαπραγματεύσει για τη Συμφωνία περί Περιβαλλοντικών Αγαθών. Με τη, συμφωνία αυτή θα μειωθούν οι δασμοί 45 ε, περιβαλλοντικών αγαθών που οι ηγέτες του ΕΠΕΚ ε, συμφώνησαν να μειώσουν τους δασμούς και στη συνέχεια θα ε, επεκταθεί αυτό το μέτρο και στις περιβαλλοντικές υπηρεσίες. Θεωρούμε ότι χρειάζονται περισσότερα μέτρα για να επιταχυθούν οι διαπραγματεύσεις αυτής της συμφωνίας και να εγκριθεί προκειμένου να τηρηθεί και η συμφωνία των Παρισίων αλλά και η αναπτυξιακή στόχη της χιλιετίας των Ηνωμένων Αθηνών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 untuk mengubah limbah menjadi energi juga dilaksanakan untuk mendukung ekonomi yang bersifat regeneratif. Thank you. The last point that I would like... Και το τελευταίο σημείο που θα ήθελα να αναφέρω αφορά την κυκλική οικονομία. Η κυβέρνηση της Ινδονησίας προωθεί αυτή τη στιγμή τη μετάβαση από την γραμμική στην κυκλική οικονομία, ώστε να αξιοποιήσουμε τους φυσικούς πόρους, τονώνοντας την, εθνική, την οικονομική ανάπτυξη. Και μάλιστα πολιτικές για τη διαχείριση των στερεών απορριμμάτων ήδη υπάρχει, ε, καθώς και δημιουργία ε, σταθμών παραγωγής ηλεκτρισμού στις χωματερές, ώστε να έχουμε μία ε, οικονομία που θα αυτοαναζωογονείται. Ευχαριστώ. Thank you, Ευχαριστώ. Αξιότιμη βουλευτά από την Ινδονησία για την παρέμβασή σας. Ε, είχαμε πάρα πολύ θετικές ιδέες. Ε, θα μπορούσαμε να τις ε, υιοθετήσουμε και ξέρω ότι θίξατε και το θέμα του φινικελαίου που είναι ένα επίμαχο ζήτημα. Έχουν υπάρξει κάποιες επίμαχες συζητήσεις μεταξύ μόνο της Ινδονησίας και της Μαλαισίας. Και πιστεύω ότι έχουμε καταλήξει σε ένα συμβιβασμό που ουσιαστικά διασκεδάζει αρκετού από του φόβου σα. Οι βουλευτέ ε, έχουν επισκεφτεί ε, και έχουν δει κάποιες από τις προκλήσεις. Όμως, αναρωτιέμαι αν κάποιος από τους εμπειρογνώμονες θα ήθελε να απαντήσει σε κάποιες από τις ε, ιδέες που ακούστηκαν σε ό,τι αφορά πρέπει το σχάρι το αυξανόμενο εμπόριο σε περιβαλλοντικά αγαθά. Αν έχουμε κάτι σχετικά, θέλετε να σχολιάσετε ή να προχωρήσουμε. Ε, από εσά εξαρτάται. Είχαμε πολλές ενδιαφέρουσες ιδέες και θα ήθελα να επανέλθω σε ένα άλλο θέμα που έθεσε ο συνάδελφος από την Ορβηγία για τα πλαστικά και ίσως ε, θα επανέλθουμε και θα έχουμε μια συζήτηση γι' αυτό όταν ε, θα έχουν όλοι ολοκληρώσει τις παρεμβάσεις τους. Έχω τώρα τον γερουσιαστή από την Ιταλία, Φριαντσέσκο Τσακομπέη. Υποθέτω ότι διαφέρει η παρέμβασή σας από την τελική παρέμβαση. Παρακαλώ, έχετε το λόγο. Ναι, είναι διαφορετική η παρέμβαση. Αυτά. Είναι αυτά που είχα σκεφτεί να πω, τα οποία ενισχύθηκαν και από αυτά που ακούστηκαν μέχρι τώρα και δεν ε, έχουν ε, σχέση με τις προσωπικές μου απόψεις. Καταρχήν θέλω να σας ευχαριστήσω που μου δώσετε την ευκαιρία να κάνω κάποια σύντομα σχόλια. Like uh, Όπως ε, και ο φίλος μας ε, από την Κίνα είπε νωρίτερα, τα αγγλικά μου τα έμαθα και εγώ σε μια ε, αγγλόφωνη χώρα αλλά τα έμαθα σε αγγλόφωνη χώρα αφού όμως είχα κλείσει τα 26 μου έτη έτσι λοιπόν τα μιλάω, αλλά με συσυλλική προφορά, συγκελένη προφορά. Έχω τρεις ερωτήσεις που σχετίζονται με το θέμα αυτό. Και να πω ταξί, συμφωνώ ότι η κλιματική αλλαγή δεν γνωρίζει σύνορα. Είναι μια δήλωση που έγινε στην αρχή και νομίζω ότι είναι πολύ σημαντική δήλωση αυτή. Είναι ένα κοινό πρόβλημα. Ακούσαμε τους συναδέλφους από την Ερβηγία... Όταν ε, μιλάμε για τους ωκεανούς, ε, πάρα πολλές χώρες ε, πλήττονται από το τι συμβαίνει στους ωκεανούς. Όμως ακόμη και σήμερα άκουσα κάποιες αναφορές για εθνικές δράσεις για την καταπολέμηση της μεταβολής του κλίματος και της περιβαλλοντικής μεταβολής. Όμως δεν άκουσα πολλά για κοινή προσπάθεια για κάποια προγράμματα, κάποια project όμορων χωρών. Γιατί εφόσον λέμε ότι είναι κοινό το πρόβλημα, θα ήταν καλό να συνεργαστούν και γειτονικέ χώρε. Μήπω θα πρέπει να ενθαρρύνουμε λοιπόν κοινά συντονισμένα project μεταξύ γειτονικών χωρών. Η δεύτερη ερώτησή μου έχει να κάνει με το τι έχει γίνει μέχρι τώρα. Και ως μέλος ε, του Τελικού Κοινοβουλίου Δηλώνω ικανοποιημένο με το γεγονό ότι η Ιταλία έχει επικυρώσει το πρωτόκολλο του Κιώτο, έχει εργαστεί προ την επίτευξη των στόχων, έχει πετύχει κάποιο από αυτού και προσπαθεί να σεβαστεί και του στόχου των Παρισίων για το 2020. Αλλά αναρωτιέμαι και για την εταιρική κοινότητα τι έχει αλλάξει στην προσέγγιση τη κοινότητα προ την ε, κλιματική αλλαγή. Τι έχουμε κάνει για να ενημερώσουμε όλο τον πληθυσμό, την κοινότητα, ότι οι καθημερινές δράσεις μας μπορεί να έχουν αρνητική ή θετική επίπτωση στην επίτευξη των στόχων τουλάχιστον δεν είναι ένα στόχο που θέλουμε να πετύχουμε μέσω μια αθλητική εκδήλωση, αλλά ε, στοχεύει στο να γίνει ο κόσμο καλύτερο για να ζούμε. Τι μπορούμε να κάνουμε για να ενθαρρύνουμε τι κοινότητέ μα, λοιπόν, να συμμετέχουν σε αυτά τα γενικά προγράμματα. Και ε, νομίζω ότι ε, θα πρέπει να αναλάβουμε και άλλες δράσεις ε, πέρα από τις εκστρατείες που έχουμε τώρα για συμμετέχει Το τρίτο είναι το, η επίπτωση στην οικονομία. Το θέμα μας σήμερα. Η κλιματική αλλαγή, κατά την άποψή μου, παράγει πολλές οικονομικές ευκαιρίες και πιθανά ωφέλη. Ακούσαμε σήμερα πολλές χώρες μια μεγάλη ζήτηση για τεχνολογίες φιλικές προς το περιβάλλον, για προγράμματα συνεργασίας, στο να, πώς θα αναπτυχθούν ε, τρόποι επενδύσεων για να έχουμε καλύτερη γη, για καλλιέργειες, πώς μπορούμε να έχουμε μηχανήματα που να λειτουργούν διαφορετικά από τα μηχανήματα που έχουμε χρησιμοποιήσει μέχρι τώρα. Αυτό και από μόνο το αποτελεί μια ευκαιρία, κυρίως για τις αναπτυγμένες, αναπτυσσόμενες χώρες, συγγνώμη, αλλά και για χώρες ε, όπως η Ιταλία που καφιέται ότι είναι μία από τις κορυφαίες χώρες του κόσμου που παράγει μηχανήματα που χρησιμοποιούνται παγκοσμίω. Αναρωτιέμαι λοιπόν τι έχουμε κάνει μέχρι τώρα και τι θα πρέπει να κάνουμε εμείς ως ε, ε, νομοθέτες, ε, ως χαράκτες της πολιτικής. Εμείς θα συνεισφέρουμε στο να αναπτύξουμε πολιτικές που θα εφαρμοστούν και θα εκτελεστούν στη συνέχεια από τις κυβερνήσεις. Τι περισσότερο μπορούμε να κάνουμε λοιπόν έτσι ώστε σε αυτά τα μεγάλα έργα να εμπλέξουμε και τις μεγάλες επιχειρήσεις να επενδύσουν με τέτοιο τρόπο έτσι ώστε το αποτέλεσμα να βοηθήσει όχι μόνο τις χώρες μας αλλά είναι και πιο φιλικές προς το περιβάλλον αλλά να επενδύσουν και στις χώρες όπου δεν ε, υπάρχει η τεχνολογία και απαιτείται η τεχνολογία αυτή για να μπορέσουμε να εκμεταλλευτούμε αυτές τις οικονομικές ευκαιρίες. Και το τελευταίο μου σχόλιο είναι ότι τίποτα που θα κάνουμε δεν θα είναι αποτελεσματικό αν δεν δράσουμε στις χώρες που ζητούν βοήθεια και έχουν πληγεί περισσότερο. Έχουμε και μεταναστευτικά ζητήματα που συζητούνται στην άλλη ομάδα. Αυτό σχετίζεται με τις ε, περιβαλλοντικές καταστροφές. Και αυτό είναι ένα μεγάλο ζήτημα και δεν μπορούμε να το γνωρίσουμε ως μέρος της οικονομικής μας ανάλυσης. Αν όσα κάνουμε στις χώρες όπου έχουμε την ευτυχία να είμαστε πιο προηγμένοι τεχνολογικά και πιο αναπτυγμένοι και μπορούμε να κάνουμε τα πράγματα καλύτερα. Αν εμείς λοιπόν δεν μεταφέρουμε τη δράση μας στις χώρες όπου πράγματι χρειάζεται, τότε όχι μόνο δεν θα πετύχουμε οικονομική ανάπτυξη, αλλά θα έχουμε ε, ουσιαστικά συνέπειες όπως βλέπουμε μετανάστευση ολόκληρων πληθυσμών. Σας ευχαριστώ. Ευχαριστώ πολύ. Πάρα πολλά μας είπατε που μας προβληματίζουν. Για να απαντήσω στο πρώτο σας σχόλιο, θα πρέπει να μιλήσουμε περισσότερο για κοινέ δράσεις μεταξύ όμορων χωρών πριν ε, λίγε εβδομάδες ε, πήρα θάρρος γιατί είχα πάει στο ε, Ασιατικό Κοινοβουλευτικό Φόρουμ και για πρώτη φορά ένιωσα ότι όλοι οι βουλευτές από τις 10 ασιατικές χώρες μιλούσαν για την αλλαγή του κλίματος με παρόμοιο τρόπο. Στο Κοινοβουλευτικό Φόρουμ του ΑΣΕΑΝ. Και ε, νομίζω ότι μπορούμε να έχουμε περισσότερα project. Μιλήσαμε για το Φινικέλαιο. Το Φινικέλαιο δεν, ε, δεν αφορά μόνο την Ινδονησία, αλλά και τη Μαλαισία. Και έχει αντίκτυπο όλη την ατμόσφαιρα και στο περιβάλλον ε, στην Νοτιοανατολική Ασία. Έτσι λοιπόν, ό,τι και να κάνει, θα πρέπει να ενέχει όλε τι όμορφε χώρε. Είναι σημαντικό κάτι τέτοιο γιατί πιστεύω ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση ε, ουσιαστικά είναι ένα project που έχει αναγνωρίσει ότι ε, πολλά πράγματα τα κάνουμε από κοινού και έχουμε και project διατομεακά. Εγώ εργάζομαι για τα βιώσιμα οικονομικά αυτή τη στιγμή, την εφόρο οικονομία, αλλά ξέρω ότι οι συνάδελφοι εργάζονται επί της κυκλικής οικονομίας ή εργάζονται στον τομέα των ε, βιώσιμων μεταφορών. Ξέρω ότι συνεχίζονται οι εργασίες εδώ, αλλά θα ήθελα να στραφώ στον κύριο Νάτπιλ και να ρωτήσω, υπάρχουν κάποια project που θα μπορούσατε να μας αναφέρετε. Και το τρίτο σημείο για τις σημαντικές ευκαιρίες που προσφέρονται στις αναπτυσσόμενες χώρες. Και τι μπορούμε να κάνουμε εμείς, τι πρέπει να κάνουμε ως ε, χαρακτής πολιτικής. Ίσως ε, και συνάδελφος από τη Ρουμανία θα ήθελε να αναφερθεί στο τι μπορούμε να κάνουμε για να ενημερώσουμε περισσότερο τους πολίτες, ε, να στείλουμε αυτά τα μηνύματα στους πολίτες. Και τα σχόλια που έκανε ο κυρίος Γερουσιαστής. Πρέπει να απευθυνθούμε στις ε, χώρες που έχουν πληγεί περισσότερες και ε, θα ήθελα να στραφώ σε εσά, γιατί είστε μία από τι χώρε που έχετε πληγεί περισσότερο, να μας δώσετε κάποιες προτάσεις για το πώς ε, θα κινηθούμε. Κάνατε κάποιες προτάσεις προηγουμένως, αλλά ίσως να έχετε και κάτι να προσθέσετε. Ποιο θέλει να ξεκινήσει, οποιοδήποτε. Για το ζήτημα της ε, υποστήριξης έργων επιτόπου, θέλω να επαναλάβω την έκκλησή μου οι ανεπτυγμένες χώρες να ξεκινήσουν το δεύτερο γύρο ε, δεσμεύσεων για το Ταμείο Πράσινου Κλίματος. Ίσως μπορεί να ξεκινήσει αυτή τη διαδικασία η κυβέρνηση της Ιταλίας. Πρέπει να τη συγχαρούμε για το γεγονός ότι είναι μία από τις πρώτες χώρες που ανακοίνωσε τη σταδιακή κατάργηση του, του άνθρακα στο 2025 και είναι και μία από τις πρώτες χώρες που ε, ανέλαβε δεσμεύσεις ε, το 2014 για τη χρηματοδότηση του Ταμείου για το Πράσινο Κλίμα. Ίσως λοιπόν μπορεί να δώσει το καλό παράδειγμα. Υπάρχουν μια σειρά από έργα που προέρχονται από αναπτυσσόμενες χώρες που ζητούν χρηματοδότηση από το Ταμείο. Δυστυχώς ε, βεβαίως υπάρχουν προβλήματα, υπάρχουν πολλές βελτιώσεις που μπορούν και πρέπει να γίνουν. Όμως Μεταξύ αυτών ε, πρέπει να σας πω ότι έχουμε λάβει πολύ ε, ενδιαφέροντα ε, προγράμματα για χρηματοδότηση από το Ταμείο. Βεβαίως υπάρχει μια συσσόρευση και μια στενοπός πρέπει να επιταχυνθούν οι διαδικασίες γιατί πολλές φορές χρειάζονται μέχρι και δύο χρόνια για να ξεκινήσει η χρηματοδότηση. Παρόλα αυτά, το ταμείο αυτό εξακολουθεί να είναι τον βασικό, είναι ο βασικός χρηματοδοτικός βραχίωνας της συμφωνίας πλαίσιο του ΟΗΕ. Αν αποτύχουμε με αυτό, με αυτό το ταμείο δυστυχώς φοβάμαι ότι δεν θα έχουμε πολλές ε, άλλες ευκαιρίες για να υλοποιήσουμε και να χρηματοδοτήσουμε έργα για την αντιμετώπιση κλιματικής αλλαγής. Θέλω να απαντήσω και εγώ στον Ιταλό συνάδελφο και σε ορισμένα ερωτήματα που έθεσε και η Πρόεδρος. Πρώτα απ' όλα θα ήθελα να πω το εξής. Η κλιματική αλλαγή είναι διαφορετική και αντιμετωπίζουμε διαφορετικές προκλήσεις, διαφορετικές ανάγκες στα διάφορα μέρη του κόσμου. Εγώ προέρχομαι από εύκρατη χώρα και μάλλον ε, χρειάστηκε περισσότερος χρόνος έως ότου και εμείς στη δική μου χώρα να συνειδητοποιήσουμε το μέγεθος του προβλήματος γιατί υπήρχαν ε, φέτος για παράδειγμα προβλήματα τα οποία δεν είχαμε ξανά αντιμετωπίσει πλημμύρες, ξηρασία και μάλιστα ε, πολύ κοντά το ένα χρονικά μετά Αντιμετωπίζουμε λοιπόν ακραία καιρικά φαινόμενα, ακραίες ε, καιρικέ συνθήκες που πλήττουν σοβαρότατα και την οικονομία μας. Αλλά δεδομένου ότι οι ανάγκες και οι προκλήσεις που αντιμετωπίζουμε ε, είναι διαφορετικές, παρόλα αυτά πρέπει να βρούμε το κοινό έδαφος. Και αυτό είναι ακριβώς που θεωρώ εγώ ότι είναι σημαντικό σε πολιτικό επίπεδο γιατί όταν μιλούμε για σταδιακή κατάργηση της χρήσης του άνθρακα ένα βασικό στοιχείο που χρειαζόμαστε είναι το θάρρος γιατί ψυχολογικά προβάλλεται αντίσταση στην αλλαγή και αυτό είναι πολύ φυσιολογικό σε κάθε αλλαγή ε, υπάρχει μια αντίσταση άλλωστε οι αλλαγές αυτές δεν είναι καθόλου εύκολες και θα είναι και δαπανηρές το θετικό όμω είναι, επανερχόμενος στην τεχνολογία, είναι το γεγονό ότι οι αλλαγέ αυτέ είναι πλέον οικονομικά προσιτέ. Δεν είναι τα πράγματα όπω ήταν πριν από κάποια χρόνια. Λίγα ε, όπου οι τεχνολογίε αυτέ βρίσκονταν ακόμα σε δοκιμαστικό στάδιο. Πλέον υπάρχουν πραγματικέ τεχνολογικέ εφαρμογέ στην αγορά και πλέον είναι οικονομικό προσιτό, είναι οικονομικά εφικτό να αξιοποιήσει τι νέε τεχνολογίε. Για τα συνεργατικά ε, project μεταξύ όμορων χωρών. Νομίζω ότι αυτό είναι ένα ε, επόμενο στάδιο στο οποίο πρέπει να περάσουμε. Είναι κάτι που είναι σύνηθες στην Ευρώπη ε, να μιλούμε για την ενεργειακή ασφάλεια και, την ενεργεια... και τις ενεργειακές αγορές. Γιατί αυτός είναι ένας από τους βασικούς μας φόβους που μας ε, αναγκάζει και μας οδηγεί στο να συνεχίζουμε να χρησιμοποιούμε ορυκτά καύσιμα. Άπαξ και ενοποιήσουμε τις, ε, τους πόρους μας, τις δυνάμεις μας και διασφαλίσουμε την ενεργειακή μας ασφάλεια, νομίζω ότι θα είναι πολύ πιο εύκολο να περάσουμε σε μια ε, οικονομία πλήρως απαλλαγμένη από τον άνθρακα και νομίζω ότι αυτή είναι η πορεία που πρέπει να ακολουθήσουμε. Επίσης, μου άρεσε πολύ το σχόλιο αυτό για το γεγονός ε, αυτό που υπόθηκε ότι η κλιματική αλλαγή είναι και ευκαιρία και να αναφερθώ και σε αυτό που είπε ο συνάδελφος από την Νορβηγία για τους ωκεανούς. Εγώ θέλω να εστιάσω στο ότι η τεχνολογία και το θάρρος είναι δύο στοιχεία που χρειαζόμαστε για το μέλλον. Και υπάρχει εδώ ένα έργο για την ε, καλλιέργεια φυκιών στη θάλασσα. Θα μπορούσαν τα φύκια να αποτελέσουν σημαντική πηγή τροφίμων Ταυτόχρονα όμως μπορούν να αποτελέσουν και έναν πνεύμονα των ωκεανών μας για, τον, για την απαλλαγή της ατμόσφαιρας από την περίσσια διοξιδίου του άνθρακα. Να για παράδειγμα, οικονομικά προσωπικές αλλαγές που υπάρχουν παραδείγματα τα οποία πρέπει να συζητήσουμε μαζί, διότι κάποιες φορές υπάρχουν λύσεις που ενδέχεται να είναι κατάλληλες ή ενδεδειγμένες για ένα μέρος του, του, του πλανήτη, αλλά όχι για άλλα μέρη του πλανήτη. Εμείς, για παράδειγμα, δεν έχουμε πρόσβαση σε ωκεανούς, έχουμε όμως άλλα ε, μέσα, όπως για παράδειγμα έχουμε αρχαίγωνα δάση και μάλιστα σε πολύ μεγαλύτερο βαθμό από ότι άλλες ευρωπαϊκές χώρες τα οποία μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε για την αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής τέτοια παραδείγματα ενώ τα οποία μπορούμε να συζητήσουμε μπορεί να διαφέρουν τα παραδείγματα, τα παραδείγματα ε, ή οι λύσεις που θα προκριθούν σε κάθε χώρα αλλά έχοντας κατά νου ότι τα προβλήματα αυτά μας αφορούν όλους νομίζω ότι είναι ένα στοιχείο το οποίο μπορεί να διευκολύνει τη συζήτηση αυτή. Θα ήθελα να απαντήσω στο ερώτημα πώς οι αναπτυσσόμενες χώρες μπορούν, ε, πώς οι ανεπτυγμένες χώρες μπορούν να βοηθήσουν τις πιο ευάλωτες χώρες. Νομίζω ότι φόρουμ σαν το σημερινό είναι ιδανική ευκαιρία για τέτοιου είδους συζητήσεις για το μέλλον και για το πώς θα δημιουργήσουμε επικοδομητικές εταιρικέ σχέσεις βοηθώντας τις ευάλωτες χώρες. Γιατί οι ανεπτυγμένες χώρες ήδη έχουν εκδηλώσει ενδιαφέρον για τέτοιες εταιρικέ σχέσεις προκειμένου να βοηθήσουν τις πιο ευάλωτες χώρες. Οπότε καλό θα ήταν να έχουμε κάποιο στρατηγικό μηχανισμό για να δημιουργήσουμε ένα πρόσφορο έδαφος για τέτοιου είδους εταιρικέ σχέσεις. Τώρα, από τη σκοπιά του Μπαγκλαντές, που είναι μία από τις πιο ευάλωτες χώρες σε ό,τι αφορά τα, τις αρνητικές συνέπειες των κλιματικών αλλαγών. Εμείς έχουμε δημιουργήσει ένα καταπιστευματικό ταμείο για τις κλιματικές αλλαγές με δικούς μας πόρους, οπότε οι ανεπτυγμένες χώρες αν ενδιαφέρονται μπορούν να συμβάλλουν σε αυτό το καταπίστευμα που έχουμε δημιουργήσει με πόρους του Μπαγκλαντές. Επίσης μπορείτε να συμμετέχετε στο επανδυτικό μας πρόγραμμα για τη δασοκομεία και τις κλιματικές αλλαγές και έχουμε και το σχέδιο ΔΕΛΤΑ για 2.100 και εκεί χρειαζόμαστε πολλές επενδύσεις και θα πρέπει να βρούμε πόρους για να το εφαρμόσουμε αποτελεσματικά. Οπότε υπάρχει, υπάρχουν πολλές δυνατότητες για συνεργασία αρκεί να εκδηλώσετε ενδιαφέρον και να λάβετε μέρος σε τέτοιου είδους επικοδομητικές εταιρικές σχέσεις. Πάνω απ' όλα όμως το πιο σημαντικό είναι η πολιτική βούληση των χωρών που θέλουν να συμμετέχουν σε τέτοιου είδους εταιρικέ σχέσεις. Σας ευχαριστώ. Λυπάμαι που άφησε τον εκπρόσωπο της Ταϊλάνδης να περιμένει τόση ώρα, αλλά ήρθε η σειρά σας επιτέλους. Σας ευχαριστώ. Κύριε και κύριοι συμπρόεδρε, αξιότιμοι καλεσμένοι, κυρίες και κύριοι, σας ευχαριστώ που μου δίνετε την ευκαιρία να σας παρουσιάσω την εμπειρία της πατρίδας μου. Είναι αναφυσβήτητο ότι οι κλιματικές αλλαγές είναι από τις μείζονες προκλήσεις για το ανθρώπινο γένος. Λόγω των ανεξέλεγκτων δυνάμεων της φύσης. Θα πρέπει να έχουμε αποτελεσματικά σχέδια και κατάλληλη εφαρμογή του σε κάθε χώρα, καθώς και συνεργασία μεταξύ των εμπλεκομένων σε όλα τα επίπεδα, προκειμένου να αντιμετωπίσουμε αυτές τις προκλήσεις. Σε εθνικό επίπεδο ε, έχουμε υπολογίσει ότι οι κλιματικές αλλαγές επηρεάζουν 1,2 δισεκατομμύρια ε, θέσεις απασχόλησης, ιδιαίτερα ε, στη γεωργία, την αλία και τη δασοκομεία. Ε, ως εκ τούτου, ο, όσοι ασχολούνται με τη διαχείριση των κλιματικών αλλαγών θα πρέπει να συνεργάζονται πιο πολύ με κοινέ και επιμερισμένες ευθύνες και κοινή διαχείριση των ικανοτήτων. Με βάση τη Συμφωνία Πλαίσιο των Ηνωμένων Εθνών για τις κλιματικές αλλαγές φάνηκε ότι είναι σημαντικό οι αναπτυγμένες χώρες να πρωτοστατήσουν στη μείωση των εκπομπών διοξιδίου του άνθρακα και να βοηθήσουν τις αναπτυσσόμενες χώρες ή τις λιγότερα αναπτυγμένες χώρες με το καλό τους παράδειγμα. Κυρίες και κύριοι, Λόγω γεωγραφικών συνθηκών και του τροπικού κλίματος, η Ταϊλάνδη έχει εδώ και δεκαετίες ε, αντιμετωπίσει τις συνέπειες των κλιματικών αλλαγών. Ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα είχαμε το 2011, όπου είχαμε στην Ταϊλάνδη τις χειρότερες πλημμύρες των τελευταίων 50 χρόνων. Πάνω από τα δύο τρίτα της χώρας πλημμύρισαν και είχαμε σοβαρότατες ζημίες στην οικονομία μας λόγω αυτών των εκτεταμένων πλημμυρών και ζημίες στην κοινωνία και τη βιομηχανία μας. Πολλά εργοστάσια χρειάστηκε να κλείσουν με αποτέλεσμα την αύξηση της ανεργίας. Και η Παγκόσμια Τράπεζα υπολόγισε τις ε, ζημίες μας σε 44 δισεκατομμύρια δολάρια. Σοβαρό πλήγμα για την ταϊλανδέζικη οικονομία και την εμπιστοσύνη που είχε παγκοσμίω. Γι' αυτό και το θέμα αυτό συμπεριλήφθηκε στο ε, σχέδιο εθνικής οικονομίας και κοινωνικο ανάπτυξης. Και από το 2012 και τα τελευταία χρόνια με το εθνικό μας στρατηγικό σχέδιο προσπαθήσαμε να βελτιώσουμε την ενημέρωση και τη συνειδητοποίηση των συνεπειών των κλιματικών αλλαγών, της ανάγκης μετριασμού των αλλαγών και προσαρμογής στις αλλαγές. Θα πρέπει να ενισχύσουμε τις ικανότητές μας να αντιμετωπίσουμε τις κλιματικές αλλαγές στους πιο ευάλωτους κλάδους, όπως είναι η δάτινη πόρη και η διαχείριση των αποβλήτων, η γεωργία και η ασφάλεια. Μόνο έτσι θα μετριάσουμε τις συνέπειες των κλιματικών αλλαγών. Και εμείς ως κοινοβουλευτικοί θα πρέπει να συνεργαστούμε στενά με τη διοίκηση και την κυβέρνηση και να βρούμε αποτελεσματικούς τρόπους για να αντιμετωπίσουμε τις παγκόσμιες προκλήσεις. Θέλουμε αποτελεσματικά νομοθετικά μέτρα οι νόμοι και οι κανονισμοί δεν θα πρέπει να είναι μόνο επίκαιροι, αλλά να εφαρμόζονται και ε, συνεκτικά και αποτελεσματικά. Και λαμβάνοντας υπόψη τον οικονομικό αντίκτυπο των κλιματικών αλλαγών, ε, στην Ταϊλάνδη χρειάστηκε να αναθεωρήσουμε πολλά νομοθετικά μέτρα και να εγκρίνουμε πολλά ε, πολλές νομοθετικές δέσμες μέτρων. Επίσης, ακυρώσαμε τη Συμφωνία των Παρισίων και υιοθετήσαμε νομοσχέδια για την καλύτερη περιβαλλοντική διαχείριση και την ε, καλύτερη ενεργειακή πολιτική και πολιτική διαχείριση αποβλήτων. Όλες αυτές οι δράσεις ε, εξασφαλίζουν κατάλληλο νομοθετικό πλαίσιο ώστε να μπορέσει η κυβέρνησή μας να αντιμετωπίσει τα προβλήματα αποτελεσματικά. Και λόγω των σοβαρών πλημμυρών το 2011 η Ταϊλάνδη αποδίδει όλο και μεγαλύτερη προσοχή στις κλιματικές αλλαγές και τα συνεφή ζητήματα. Και αυτή την προσοχή τη δίνουν όχι μόνο ο δημόσιο και ιδιωτικό τομέα, αλλά και οι ιδιώτε που θα πρέπει να λάβουν υπόψη τι κλιματικέ αλλαγέ. Κάτι τέτοιο προποθέτει μεγάλη υποστήριξη όλων των εμπλεκομένων φορέων, συνεργασία και δράση, προκειμένου ο πλανήτης μας να είναι ένα καλύτερο μέλος για να διαβίουμε εμείς, αλλά και οι επερχόμενες γενναίες. Ευχαριστώ. Σας ευχαριστώ. Ευχαριστώ τον εκπρόσωπο της Ταϊλάνδης. Ε, χαιρετίζω τη δήλωσή σας και επειδή ο χρόνος μας πιέζει να περάσουμε αμέσως στις Φιλιππίνες γιατί περιμένουν το Μπρουνέι, το Βιετνάμ και η Κύπρος στον κατάλογο των αγορητών. Δεν βλέπω άλλον, οπότε ολοκληρώνω το κατάλογο και θα δώσω το λόγο στις Φιλιππίνες. Σας θέλω παρακαλώ να είστε σύντομος όμως. Ευχαριστώ. Έχω μια ερώτηση μόνο κυρία Πρόεδρε. Δόθηκε τουλάχιστον από, δύο, από τους δύο κεντρικούς ομιλητές ιδιαίτερη έμφαση στη σημασία ε, της χρηματοδότησης ε, για την αντιμετώπιση των κλιματικών αλλαγών, κυρίως στις ασιατικέ χώρες. Είπατε ότι είναι απαραίτητο κάτι τέτοιο. Και μάλιστα το πιο σημαντικό έγγραφο της 10 η ΑΣΕΠ είναι το αυριανό μας ψήφισμα. Και διορθώστε με αν κάνω λάθο, αλλά έχω την αίσθηση ότι η διακήρυξη που θα υιοθετήσουμε αύριο δεν αναφέρει ιδιαίτερα τη χρηματοδότηση για το μετριασμό των κλιματικών αλλαγών. Οπότε ρωτώ του κεντρικού μα ομιλητέ, εσεί θα συστήνατε θερμά η αυριανή μα διακήρυξη να περιλαμβάνει και ρητή μνήμα τη χρηματοδότηση, ανάγκη χρηματοδότηση ε, τη αντιμετώπιση των κλιματικών αλλαγών. Γιατί το σχέδιο τη διακήρυξη έχει μόνο μία παράγραφο που ίσω σχετίζεται κάπω με το οικονομικό. Μόνο η παράγραφο 26 κάνει μία έμεση μνήμα τη χρηματοδότηση των κλιματικών αλλαγών. Ερωτώ λοιπόν τους κεντρικούς ομιλητές, είναι αρκετή αυτή η έκκληση προς τις κυβερνήσεις και τους διεθνούς δωρητές να συντονίσουν τις αναπτυξιακές πολιτικές και τις εμπορικές συμφωνίες και διατάξεις με μηχανισμούς πρόληψης των κλιματικών αλλαγών με βάση τους, τις αρχές και τις διατάξεις της Συμφωνίας των Παρισίων. Αρκεί αυτό για να καλύψουμε παρκώς το θέμα τη χρηματοδότηση του μετριασμού των κλιματικών αλλαγών. Και αν δεν είναι επαρκή αυτή η παράγραφο, δεν θα πρέπει να έχουμε και μια ρητή μνήμα της χρηματοδότηση των κλιματικών αλλαγών. Ερωτώ αν το κρίνετε σκόπιμο. Δεν ξέρω αν επιτρέπεται διαδικαστικά να καταθέσουμε τροπολογίε στο σχέδιο διακήρυξη. Ερωτώ όμω, τους κεντρικού μα ομιλητέ αν πιστεύουν ότι η παράγραφος ως έχει αντιμετωπίσει επαρκώς το ζήτημα της χρηματοδότησης. Να αποσαφηνίσω υπήρχε μια ευκαιρία τροποποίησης ε, της δήλωσης πριν να ξεκινήσουν οι συναντήσεις, ε, γιατί είχε διαναμηθεί σε όλα τα μέλη. Επίσης υπήρχε σήμερα το πρωί μια συνεδρίαση ε, τελικής σύνταξης όπου καθέ αντιπρόσωπος θα μπορούσε να έχει παρέμβει και να ζητήσει να συμπεριληφθεί το αίτημά του. Τώρα, δυστυχώς, ε, όλα τα μέρη έχουν συμφωνήσει επί του κειμένου της δήλωσης. Είναι δύσκολο να πάμε πίσω τώρα και να την τροποποιήσουμε, όμως... Ε, Κατανοώ τι ανησυχίε ότι θα πρέπει να αναφέρετε με ισχυρότερους όρους τη χρηματοδότηση για την καταπολέμηση της κλιματικής αλλαγής. Ίσως αυτό θα μπορούσε να συμπεριληφθεί σε μια μελλοντική δήλωση για την επόμενη φορά. Γιατί τώρα έχουν δεχτεί όλοι την διακήρυξη και από ό,τι καταλαβαίνω είναι και στην ιστοσελίδα. Επομένως θα είναι αρκετά δύσκολο να ξανακαλέσουμε όλους τους εταίρους της ΑΣΕΠ για να τροποποιηθεί η διακήρυξη αυτή. Αν έχετε ανησυχίες λοιπόν για το θέμα αυτό, ευχαρίστω να τις σημειώσουμε και αν θέλει κάποιος στο πάνελ να κάνει ένα σχόλιο, αλλά για να κερδίσουμε χρόνο θα ήθελα να επανέλθω στον κατάλογο των ομιλητών. Σημείωσα το σχολείο σας και θα διασφαλίσω ότι οι οργανωτές θα ακούσουν αυτό που είπετε. Ένα πολύ σύντομο follow-up. Ναι, είναι αλήθεια αυτό διαδικαστικά ότι δεν μπορούμε πλέον να κάνουμε τροπολογίες αλλά να ακούσουμε τους βασικούς ομιλητές. Αν είναι απαραίτητο για το θα πρέπει να το αντιμετωπίσουμε αυτό. Μήπως να το συζητήσουμε στο τέλος, γιατί θέλω να δώσω το λόγο σε τρεις ακόμα αντιπροσωπείες και δεν μας φτάνει ο χρόνος. Θα πρότεινα λοιπόν ε, στο τέλος να κλείσουμε με μια δήλωση ή με κάποια απάντηση από όλους τους βασικούς ομιλητές για το θέμα αυτό. Θέλετε να δώσετε το λόγο στον Μπρουνέη, παρακαλώ. Θα πρέπει να προχωρήσουμε και θα ήθελα να καλέσω τον ομιλητή από τον Μπρουνέη. Παρακαλώ. Ευχαριστώ. Πρόεδρε, που δίνετε στον Προνέη το λόγο. Να ξεκινήσω παραθέτω στο Γάλλο Πρόεδρο. Το, προ, το Φρασουά Ολάν, τον πρώην Γάλλο Πρόεδρο, καταστρέφουμε τη φύση, βλάπτουμε το περιβάλλον. Θα πρέπει η ανθρωπότητα να αναλάβουν τις ευθύνες τους για το καλό των μελλοντικών γενεών. Η κλιματική αλλαγή προέρχεται από ανθρωπογενείς δραστηριότητες μέσω των εκπομπών διοξιδίου του άνθρακα και εκπομπών αερίου του θερμοκηπίου. Αυτό προέρχεται από τη χρήση των ορεικτών καυσίμων και άλλες βιομηχανικές δραστηριότητες. Το Διεθνές Πάνελ για την Κλιματική Αλλαγή λέει ότι με τη σημερινή τάση ο πλανήτης θα μπορούσε να είναι θερμότερος κατά 1,8 βαθμούς Κελσίου στο μέλλον και σε πάνω από δύο δεκαετίες θα πρέπει να μετακινηθούμε από τα αρκτά κόψιμα σε χρήση πιο καθαρής ενέργειας. Ένα άλλο θέμα έχει να κάνει με την απεριμοποίηση. Υπάρχει συνένεση ότι αυτό το θέμα θα πρέπει να συζητηθεί στην ε, ατζέντα του Ρίο 20 και να συζητηθεί και στο διακυβερνητικό πάνελ για το LDD. Επίσης, έχουμε αποψήλωση των δασών και υποβάθμιση των τροπικών δασών και αυτό οδηγεί σε αύξηση των εκπομπών κατά 20%. Επομένως, αυτό θα, θα πρέπει να αναλάβουμε δράση για να προστατεύσουμε τη βιοπικιλότητα και να αποτρέψουμε την καταστροφή. Καθώς συνεχίζονται να αυξάνονται οι παγκόσμιες εκπομπές, παρά τις δεσμεύσεις του 2015 το βλέπουμε ότι έχουμε υψηλές ε, θερμοκρασίες, αύξηση του επίπεδου των ωκεανών ε, λόγω των εκπομπών. Γίνεται πιο θερμός ο πλανήτης ε, και σε λίγο οι ωκεανοί θα καταπιούν νησιά και θα έχουμε πρόβλημα ε, ασφάλειας για πάρα πολλούς ανθρώπους, θα πρέπει να μετακινηθούν σε άλλα μέρη και φυσικά έχουμε και πρόβλημα για το μέλλον των εργαζομένων και των αλλιέων. Υπάρχει ένας συσχετισμός της κλιματικής ε, αλλαγής. Ε, η κλιματική αλλαγή οδηγεί σε υπερθέρμανση των ωκεανών, οδηγεί σε υπερβολικές βροχοπτώσεις και σε πλημμύρες. Έχουμε λοιπόν ε, πλημμύρες ε, των ε, περιοχών που βρίσκονται σε χαμηλό υψόμετρο και αυτό έχει επίπτωση σε καταστροφή των καλλιεργιών. Επίσης, βλέπουμε ότι σε κάποιες χώρες έχουμε καύσονες και αυτό καταστρέφουν και αυτό οδηγεί, συγγνώμη, σε απερίμωση και ξηρασία. Σε κάποιες χώρες γίνεται γυμνό το έδαφος, άγωνο και αυτό έχει επίπτωση στην ασφάλεια των τροφίμων. Το Μπρουνέι Ντερεσαλάμ ήταν μέρος ε, της ε, συμφωνίας του ΙΕ, FCC, της συμφωνίας πλαίσιο για την κλιματική αλλαγή προσχωρήσαμε στο πρωτόκολλο του ΟΗΕ, FCC, το 2008. Είμαστε μια αναπτυσσόμενη χώρα. Δεν έχουμε νομικά δεσμευτικούς όρους στο πρωτόκολλο για τη μείωση των εκπομπών. Οι εκπομπές μας είναι 0,07% των ε, συνολικών εκπομπών παγκοσμίω ετησίω. Το Μπρουνέι πιστεύει ότι θα πρέπει και αυτό να εργαστεί κατά της υπερθέρμανσης του πλανήτη. Επομένως, το Μπρουνέι προσχώρησε στη Συμφωνία των Παρισίων που υπογράφηκε το 2015 και επικαιρώθηκε το Σεπτέμβριο του 2016. Θέλουμε για την καταπολέμηση της, της κλιματικής αλλαγής να αναπτύξουμε διάφορα φωτοβολταϊκά συστήματα η γίνονται φιλόδοξες επενδύσεις στην πετρελαϊκή βιομηχανία και στη βιομηχανία αερίου. Επενδύσεις της τάξης του 30%, μείωση του 30% των εκπομπών μέχρι το 2021. Έχουμε μείωση στην κατανάλωση ενέργειας και θέλουμε να φτάσουμε στα επίπεδα του 2009 μέχρι το 2030. Ε, μέχρι το 2035 θέλουμε να έχουμε τη χρήση ανανεώσιμων πηγών ενέργειας ε, στο επίπεδο του 10%. Και το Μπρουνέι συνεργάζεται με την Ιαπωνία για ένα project ε, παροχής ενέργειας από υδρογόνο. Έχουμε και ένα σχέδιο επίδειξης που θα αρχίσει να λειτουργεί τον ξεκίνησε να λειτουργεί τον Απρίλιο του 2018. Το Μπρουνέι μαζί με την Ινδονησία επικεντρώνεται στην διατήρηση των δασών και στην προστασία του οικοσυστήματος για την προστασία του περιβάλλοντος. Σας ευχαριστώ. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ε, να προχωρήσουμε σιγά σιγά προς το τέλος της συζήτησής μας. Θα ήθελα να δώσω το λόγο στον ε, εκπρόσωπο του Βιετνάμ. Συστηθείτε παρακαλώ επίσης. Ευχαριστώ. Αγαπητοί συμπροέδροι, αγαπητοί βουλευτές, Αγαπητοί προσκεκλημένοι, σας ευχαριστώ που δίνετε στην την αντιπροσωπεία τη δυνατότητα να τοποθετηθεί. Εγώ είμαι πρόεδρος της Επιτροπής ε, Παιδείας και Επιστημών της Εθνοσυνέλευσης του Βιετνάμ και θέλω να παρέμβω στην σημερινή μας συζήτηση. Όπως γνωρίζετε, το Βιετνάμ είναι μεταξύ των χωρών που έχουν πληγεί σοβαρότατα από την κλιματική αλλαγή. με βάση τον ε, δείκτη CCVI για την, ε, για την ε, ευαλωτότητα στην κλιματική αλλαγή. Η, το Βιετνάμ είναι μία από τις πιο ευάλωτες χώρες. Πάνω από 200 φυσικές καταστροφές έχουμε ζήσει τα τελευταία χρόνια. Έχουμε δυστυχώς υποστεί ε, αρνητικές επιπτώσεις και στο ΑΕΠ μας λόγω της κλιματικής ε, αλλαγής. 5%, 11% ε, του, του πληθυσμού έχει πληγεί, 7% των γεωργικών δραστηριοτήτων μας και έχουμε υποστεί μια μείωση 10% περίπου του ΑΕΠ μας λόγω των επιπτώσεων της κλιματικής αλλαγής. Λόγω της σοβαρότητας αυτής της παγκόσμιας το Βιετνάμ συμμετέχει ενεργά στις ε, διεθνείς συνδιασκέψεις και στα μέτρα που λαμβάνονται σε διεθνέ επίπεδο για την αντιμετώπιση τη κλιματική αλλαγή. Για τη βελτίωση των ε, νομικών, του, του νομικού συστήματος, τη μείωση των εκπομπών ε, αερίων του θερμοκηπίου και απαγόρευση ε, μια σειρά προϊόντων όπω είναι οι πλαστικέ σακούλες και μείωση της χρήσης ορυκτών καυσίμων. Επίσης δίνουμε κίνητρα ε, σε φιλικές προ το, προς το περιβάλλον πολιτικές και μέτρα. Η κλιματική αλλαγή δυστυχώς ε, συμβαίνει πιο γρήγορα από ό,τι περιμέναμε. Και αυτό είναι μια νέα διάσταση που απαιτεί ανάληψη δράσης και επιβολή μέτρων διαπιστώνουμε ότι οι μηχανισμοί μας δεν είναι αρκετά αποτελεσματικοί. Also uh, Um, για να ενισχυθεί λοιπόν ο συντονισμό στον, ε, στο πλαίσιο του ΑΣΕΠ για να εξυπηρετηθούν οι στόχοι του, του Παρισιού το Βιετνάμ θέλει να υποβάλει δύο προτάσεις. Πρώτον, να δημιουργηθεί και να ε, προωθηθεί ένας μηχανισμός της ΑΣΕΠ με έναν πιο απτό τρόπο μια ομάδα δηλαδή η οποία θα εξετάζει συγκεκριμένα θέματα και θα συναπαρτίζεται από εκπροσώπους Ευρώπης και της Ασίας. Μπορούμε να, ε, για παράδειγμα να εκπονούμε ε, μελέτες αντικτύπου, να διευκολύνουμε την μεταφορά τεχνολογίας, ε, την, τις συμπράξεις δημοσίου και ιδιωτικού τομέα, και διενέργεια περιβαλλοντικών ελέγχων. Οι έλεγχοι αυτοί μπορούν να ενισχύσουν την χάραξη και την υλοποίηση περιβαλλοντικής πολιτικής που θα αντιμετωπίζει την κλιματική αλλαγή. Όσον αφορά τους διδάτινους πόρους, επικεντρωνόμαστε σε προγράμματα ε, διασυνεριακής συνεργασίας για την καλύτερη διαχείριση των υδάτινων πόρων για την εξάλληψη των αρνητικών επιπτώσεων της ε, κλιματικής αλλαγής στους υδάτινους πόρους, στους πληθυσ... των αρνητικών επιπτώσεων αυτής στους πληθυσμούς που ζουν ε, κατά μήκο ε, ποταμών αλλά και σε παράκτιες περιοχές. Δεύτερον, θέλουμε να κινητοποιήσουμε και τη χρηματοδότηση, ιδίως από διεθνείς πηγές ε, για να μπορέσουμε να ανταποκριθούμε σε όλα αυτά τα μέτρα που σας περιέγραψα. Ευχαριστώ. Σας ευχαριστούμε. Και τελευταίος αλλά εξίσου σημαντικός ε, είναι ο εκπρόσωπος της Κύπρου. Παρακαλώ πείτε μας το όνομά σας. Είμαι ο Νίκος Τορναρίτης, είμαι αναπληρωτής πρόεδρος της Επιτροπής Εξωτερικών του Κυπριακού Κοινοβουλίου και την ίδια ώρα είμαι πρόεδρος της Επιτροπής Οικονομίας και Βιώσιμης Ανάπτυξης των Ασιατικών Κοινοβουλίων. Ε, το λέγω αυτό για να τονίσω τον κομβικό ε, ρόλο και γεωγραφική ειδικότερα θέση της Κύπρου, η οποία ουσιαστικά βρίσκεται στο ανατολικό άκρο της Ευρωπαϊκής Ένωσης και βεβαίως είναι πλήρες μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης και την ίδια ώρα ε, δίπλα ακριβώς από την Ασία. Πολιτικά η Κύπρος ανήκει στην Ευρωπαϊκή Ένωση, γεωγραφικά ανήκει στην Ασία. Το πρώτο που θέλω να πω είναι ότι ε, συμφωνούμε με αυτό που ακούστηκε αμέσως προηγούμενα από τον εκπρόσωπο του Βιετνάμ ότι πρέπει να δημιουργηθεί μια βάση, ένας μηχανισμός Ευρώπης Ασίας που να ασχολείται με τα θέματα του περιβάλλοντος που ίσως είναι το κρισιμότερο θέμα που απασχολεί σήμερα την ανθρωπότητα και αν θέλετε η Κύπρος είναι έτοιμη και λόγω της θέσης που σας περιέγραψα προηγουμένως να φιλοξενήσει το συγκεκριμένο μηχανισμό, τη συγκεκριμένη γραμματεία. Θα πω ότι είναι πολύ σημαντική η σημερινή και η αυριανή μέρα, γιατί φέρνει κοντά ανθρώπους από διαφορετικές χώρες, διαφορετικούς πολιτισμούς και και τους δίδει τη δυνατότητα να ανταλλάξουν σκέψεις, ε, εμπειρίες, τεχνογνωσία. Θα πω κυρίες και κύριοι, φίλες και φίλοι ότι η αηφόρα παραγωγή ενέργειας ειδικότερα ε, οι ανανεώσιμες πηγές ενέργειας κατά την άποψή μας είναι η πιο πετυχημένη στρατηγική βιώσιμης ανάπτυξης. Στην Κύπρο η ενεργειακή πολιτική είναι σύμφωνη με τους στόχους των Ηνωμένων Εθνών, με τη Συμφωνία των Παρισίων, αλλά και βεβαίως με ό,τι υποστηρίζει η Ευρωπαϊκή Ένωση όσον αφορά τη μείωση των ρηπογόνων εκπομπών και των φαινομένων που προκαλούν την υπερθέρμανση του πλανήτη και την κλιματική αλλαγή. Θέλω έτσι να είμαι σύντομος και να σας πω ότι στη χώρα μου εφαρμόζουμε ε, ε, ένα πρόγραμμα το οποίο ε, ε, μέσα από το οποίο εγκαθιστούμε ηλιακούς συλλεχτές ανακάτοικο όσον αφορά τη χρήση ηλιακής ενέργειας για θέρμανση και των οικοκυριών και των ε, επιχειρήσεων. Και η Κύπρος αυτή τη στιγμή ποσοστιαία ανακάτοικο είναι η πρώτη χώρα στον κόσμο σε ηλιακούς θερμοσύμφωνες αυτό ή αν θέλετε μέσα από αυτού μπορούμε να δώσουμε την τεχνογνωσία το πώς έχουμε πετύχει αυτόν τον συγκεκριμένο στόχο. Ενώ έχει, έχουμε σημειώσει σημαντική πρόοδο στην παραγωγή ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Ιδιαίτερα σε χώρες με υψηλό ετήσιο ποσοστό ηλιοφάνειας, το παράδειγμα μας μπορεί να συνεισφέρει στην οικιακή εξοικονόμηση ενέργειας και χρήματος Προ όφελο πρώτα και πάνω απ' όλα του περιβάλλοντος και δεύτερον του προπολογισμού της οικονομίας δηλαδή της κάθε οικογένεια ε, ξεχωριστά. κλείνοντα θα πω ότι στο πεδίο των ανανεώσιμων πηγών ενέργεια, επιβάλλεται συντονισμό των προσπαθειών μας για την πρόθεση της οικονομικής ανάπτυξης και της αηφόρου χρήσης της ενέργειας, για τη σύνδεση των ενεργειακών μας πολιτικών με τους παγκόσμιους στόχους για βιώσιμη ανάπτυξη και την καταπολέμηση της κλιματικής αλλαγής, καθώς και ειδικότερα την απομείωση των επιβλαβών για τη φύση και την ανθρωπότητα επιπτώσεων της και του οικονομικού αντίκτυπου αυτών των επιπτώσεων. Επειδή θα έχω την ευκαιρία αύριο ε, να μιλήσω και στα closing remarks, σας ευχαριστώ πολύ για την ευκαιρία που μου δώσατε. Να είστε καλά. Thank you very much. Σας ευχαριστούμε. Σας ευχαριστούμε πολύ που μας μιλήσατε για την πρόοδο που σημειώνει η Κύπρος στα θέματα αυτά. Θα πρέπει να ολοκληρώσουμε τώρα, αγαπητοί συνάδελφοι. Θα κάνω κάποια σκέψεις συμπερασματικές, αλλά έχουμε και το αναπάντητο ερώτημα των Φιλιππίνων. Αλλά να δώσω και το λόγο στους καλεσμένους μας σε ένα λεπτό αν θέλω να κάνω μια σύνοψη, να κεφαλώσουν κάτι και στο τέλος θα καλέσω και τον εισηγητή μας, τον γερουσιαστή από την Ιταλία, να κάνει μια σύντομη ανακεφαλαίωση. Θα δώσω λοιπόν ένα λεπτό στον καθένα καλεσμένο, θα πω εγώ κάποια συμπερασματικά σχόλια και μετά θα δώσω και στον εισηγητή μας το λόγο και λέγες σύντομες παρατηρήσεις. Ε, πρώτα καλεσμένη από τον Μπαγκλαντές. Ευχαριστώ. Θα ήθελα να απαντήσω στις παρατηρήσεις που κάνατε, στην πολύ σημαντική παρατήρηση που έκαναν οι Φιλιππίνες για τη χρηματοδότηση του κλίματος. Σίγουρα το θέμα αυτό είναι αναπόσπαστη και απαραίτητη συνιστόσα όλων των συζητήσεων για την καταπολέμηση των προκλήσεων που δημιουργούν οι κλιματικές αλλαγές και μια και δεν είναι δυνατόν να συμπεριληφθεί κάτι τέτοιο στη διακήρυξη της 10ης ΑΣΕΠ, θεωρώ ότι παρόλο που δεν αναφέρεται ρητά, υπάρχει εμέσω αυτό το ζήτημα στη διακήρυξη. Γιατί η διακήρυξη αναφέρεται στη Συμφωνία των Παρισίων, στη Συμφωνία Πλαίσιο των Ηνωμένων Εθνών για τις κλιματικές αλλαγές και σε άλλου μηχανισμού. Οπότε έστω και έμεσα μπορούμε να θεωρήσουμε το ζήτημα των πόρων, της διαχείρισης των πόρων, της χρηματοδότησης, του κλιματικού ταμείου υπάρχουν έστω και έμεσα στη διακήρυξη. Οπότε σε κάποιο βαθμό λαμβάνεται υπόψη αυτός ο προβληματισμός σας, παρόλο που δεν γίνεται ρητή ξεκάθαρη μνήμα. Μάλιστα, ευχαριστώ ο κύριος Άλλεν. Το περισσότερο λεπτό μου θα το αφιερώσω στην απάντηση τη ερώτηση από τι Φιλιππίνε. Φυσικά χρειαζόμαστε χρηματοδοτικά μέσα και μηχανισμού και συμμετείχα στη πρωινή συντακτική επιτροπή ε, τη διακήρυξη και σα διαβεβαιώ ότι έγιναν εκτενεί και πολύ καρποφόρε συζητήσει. Πολλά σημεία εξετάσαμε και πολλέ τροπολογίε αναλύσαμε. Ακόμη και αυτό που αναφέρατε εσεί, ότι είπατε ε, μιλήσετε για την παράγραφο 26. Έγιναν τέσσερι διαφορετικές προτάσεις για την παράγραφο 26. Θα πρέπει να δούμε τι αναφέρει στο σελίδα για την παράγραφο αυτή. Γιατί ίσως τελικά βελτιώθηκε το τελικό κείμενο της παραγράφου 26 χάρη στι τροπολογίες. Ίσως έχει περισσότερες ιδέες και μνήες και για το ζήτημα τη χρηματοδότηση. Επίση, θα ήθελα να σε επισημάνω την παράγραφο 37 και εκεί αναφέρονται τα χρηματοδοτικά μέσα και οι πηγές και απευθύνει η έκκληση στα κράτη-μέλη να συνεργαστούν για να ενισχύσουν τη χρηματοδότηση. Επίσης χρειαζόμαστε σίγουρα χρηματοδοτικά μέσα, αλλά θα πρέπει να ξεχνούμε το ευρύτερο πλαίσιο που έχουμε σήμερα, γιατί μετά την αποχώρηση μιας μεγάλης χώρας από τη Συμφωνία των Παρισίων, διατρέξαμε τον κίνδυνο να πρέπει να αναδιατυπώσουμε όλε τι δεσμεύσει. Και αυτή είναι η βασική αξία τη διακήρυξη. Το γεγονό ότι βρισκόμαστε εδώ σήμερα και όλοι επανεπιβεβαιώνουμε τι δεσμεύσει μα, να τηρήσουμε του στόχου ε, μα και να αντιμετωπίσουμε τι κλιματικέ αλλαγέ, αυτό είναι πολύ σημαντικό. Και ε, η θέση μα σήμερα είναι πολύ σημαντική, γιατί πραγματικά η διακήρυξη υπέρχει πολλά θετικά σημεία και πραγματικά είναι πολύ σημαντικό και μεγάλη επιτυχία ότι μιλούμε και για τη μετανάστευση και για άλλους παράγοντες και ανοίγουμε την προοπτική και για περαιτέρω συζητήσεις για τα χρηματοδοτικά μέσα. Τα υπόλοιπα σας τα είπε η Πρόεδρος ως προς τη διαδικασία και το αν ε, είναι δυνατή περαιτέρω υποβολή τροπολογιών. Πάντως επαναλαμβάνω την ανάγκη να δείξουμε θάρρος, τεχνολογία, να εκμεταλλευτούμε την τεχνολογία και να ενισχύσουμε τη συνεργασία μεταξύ μας. Ευχαριστώ. Θα ήθελα και εγώ να αφιερώσω το λεπτό μου σε δύο σημεία. Το πρώτο δεν ε, ε, σχολιάστηκε επαρκώς στη συζήτηση. Θα ήθελα να απευθύνω και πάλι μια επιτακτική έκκληση προς τις ασιατικές χώρες να δώσουν προτεραιότητα στη συζήτηση για τη χρήση της γης. Αυτή είναι η στρατηγική απάντηση στην προκλήση που δημιουργεί το, το κλίμα για την παραγωγή τροφίμων. Θα πρέπει να δώσουμε προτεραιότητα στην τροφή, παραγωγή τροφίμων και κυρίω για εγχώρια κατανάλωση και όχι για εξαγωγέ. Δεύτερο ζήτημα, η χρηματοδότηση του κλίματο. Λυπούμε, αλλά εγώ συμμετείχα τα τελευταία 12 χρόνια σε πολλέ διαπραγματεύσει τη διάσκεψης των μερών και μετά τη Συμφωνία των Παρισίων υπήρξε μεγάλη απροθυμία εκ μέρου των ανεπτυγμένων χωρών να υποβάλλουν συγκεκριμένες δεσμεύσεις για, τα χρημα... για τη χρηματοδότηση για να βρεθούν τα 100 δισεκατομμύρια το χρόνο που ε, αναφέρονται στην Συμφωνία των Παρισίων και στην υπόσχεση που δόθηκε εκεί. Θα πρέπει να είμαστε ε, σαφείς και ρητίως προς τις δεσμεύσεις και να υπάρχει και ένα συγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα για την υλοποίηση των υποσχέσεων για τη χρηματοδότηση του κλίματος. Μάλιστα. Και τώρα ο λόγος στον συμπρόεδρο, τον καθηγητή UN, για να πει και αυτός δύο λόγια. Θα ήθελα και εγώ να τονίσω επ' ευκαιρία το πρώτο σχόλιο του προσώπου της Ιταλίας για την ανάγκη συντονισμένων προσπαθειών. Στην Κίνα όλο και περισσότερο έχουμε συντονισμένες προσπάθειες και κοινέ ε, επιχειρήσεις και διεθνή συνεργασία. Θα σας δώσω μερικά παραδείγματα και θα ήθελα επ' ευκαιρία να ευχαριστήσω την Ιταλική κυβέρνηση γιατί το Υπουργείο Περιβάλλοντος της Ιταλίας δόρισε ένα ολόκληρο κτίριο που λειτουργεί μόνο με ηλιακή ενέργεια πριν από 7 χρόνια στη Κίνα. Και πίνος, έχουμε μια διεθνή κοινή επιχείρηση στο πανεπιστημιακό, στο ακαδημαϊκό επίπεδο και εγώ είμαι από το ε, Πανεπιστήμιο της Σανγκάης. Εκεί είχαμε τα ερευνητικά Ινστιτούτα της Τοϊότα και της Τσίνχουα στην Σανγκάη και στις αρχές του αιώνα μας το MIT από τις Ηνωμένες Πολιτείες, το Πανεπιστήμιο του Cambridge ε, από την Ηνωμένο Βασίλειο και ένα Κινέζικο Πανεπιστήμιο από κοινού έχουν συνάψει τη Συμμαχία για τη Μείωση του Άνθρακα. Επίσης ε, ιδρύσαμε ένα ε, ερευνητικό κέντρο για την περιβαλλοντική έρευνα στην Κίνα. Αυτά είναι μια, λίγα παραδείγματα του τι μπορούμε να κάνουμε και είμαι σχετικά αισιόδοξο γιατί διαπιστώνω ότι ενισχύεται η διεθνή συνεργασία και δημιουργούνται όλο και περισσότερες κοινέ επιχειρήσεις ε, παγκοσμίω. Και γι' αυτό χαιρετίζουμε κάθε μορφή έρευνας η ανάπτυξη συνεργασία στο μέλλον για τα θέματα αυτά. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ πολύ. Ακούσαμε σήμερα πολλά καλά παραδείγματα από χώρες και στην Ασία και στην Ευρώπη για την καταπολέμηση της αλλαγής του κλίματος. Θέλω να συνοψίσω κάποια σημεία προκειμένου ο εισηγητής να τα λάβει υπόψη όταν ε, θα ετοιμάσει τη δική του αναφορά για αύριο το πρωί από τις 15 μέχρι τις 10.30. Και θα ήταν καλό αν μπορούν να παρευρίσκονται και οι συνάδελφοι να τον υποστηρίξουν. Κάποια από τα κύρια μηνύματα είναι τα εξή. Πολλοί είπαν ότι οι αναπτυσσόμενε χώρε είναι οι πιο ευάλωτε σε σχέση με τον αντίκτυπο τη αλλαγή του κλίματο. Επίση, ο αντίκτυπο ε, στον τομέα τη γεωργία είναι ιδιαίτερα ανησυχητικό γιατί η πληρότητα των πολιτών στην Ασία κερδίζουν ε, το εισόδημά τους ε, από τον τομέα αυτό. Πολλοί ομιλητέ υπογράμμισαν την ιδέα τη πρόσβαση σε καθαρέ τεχνολογίε για την καταπολέμηση τη κλιματική αλλαγή. Και πιστεύω εδώ ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση μπορεί να συνεισφέρει και να μοιραστούμε την γνώση μας. Και ξέρετε, φυσικά σημειώνω και το θέμα της χρηματοδότησης ε, για την πρόσβαση σε καθαρές τεχνολογίες. Επίσης οι ομιλητές ζήτησαν να έχουμε ένα πράσινο ταμείο για το κλίμα το οποίο θα πρέπει ε, να τροφοδοτείται με κονδύλια ε, και να χρηματοδοτεί τις αναπτυσσόμενες χώρες. Αναφέρθηκαν οι ομιλητές σε πολιτικές που για την πράσινη οικονομική ανάπτυξη, όμως ε, σημείωσε και τι είπε ο γερουσιαστή από την Ιταλία, πώς μπορούμε να ενθαρρύνουμε περισσότερο τις κοινέ δράσεις μεταξύ των όμορων χωρών για την καταπολέμηση της αλλαγής του κλίματος. Και ελπίζω χώρες ε, και από το ΑΣΕΑΝ ε, μπορούν ε, να συνεργαστούν για να καταπολεμήσουν την κλιματική αλλαγή. Θέλω να επανέλθω σε μια ερώτηση που έθεσε ο βουλευτής από την Ορβηγία για το αν μπορούν να μειωθούν οι εκπομπές διοξιδίου του άνθρακα στην Ασία. Είναι σημαντικό να αντιμετωπίσουμε, να επιλύσουμε το θέμα των πλαστικών και στην Ασία και στην Ευρωπαϊκή Ένωση και την ε, μία και μόνη χρήση των πλαστικών. Δεν το συζητήσαμε αυτό, αλλά είναι πολύ σημαντικό. Νομίζω ότι χρειαζόμαστε κατάλληλη νομοθεσία για οποιαδήποτε μετατροπή, για οποιαδήποτε αλλαγή. Και φυσικά για την Ινδονησία, το θέμα του ΠΟΕ, τη ε, Συμφωνίας Περιβαλλοντικών Αγαθών και ότι χρειάζεται να ολοκληρωθούν γρήγορα οι διαπραγματεύσει. Κύριε Γερουσιαστά, θα έχετε αρκετά σημεία τα οποία θα χρειαστεί να αναφέρετε και θα ήθελα να μοιραστείτε μαζί μας οτιδήποτε άλλο σημειώσετε εσείς έτσι ώστε να ξέρουν οι συνάδελφοι αν συμφωνούν και να μπορείτε να το κάνετε και πάρα πολύ γρήγορα γιατί έχουμε και το δείπνο. Θα πρέπει οι συνάδελφοι να πάνε σε ένα άλλο κτίριο. Σας ευχαριστώ που κάνατε τη δουλειά μου, Πρόεδρε. Πολύ ωραία τα σύνοψίσατε όλα αυτά. Δεν μπορώ να προσθέσω και πολλά. Συμφωνώ απόλυτα με τα τελικά σας σχόλια και τη σύνοψη που κάνατε. Νομίζω ότι πέρα από όσα υπόθηκαν ξεκάθαρα, πολλοί ομιλητές ε, πίεσαν για την ύπαρξη συνεργατικών ε, έργων, ε, κυρίως στην ενδυνάμωση της συνεργασίας μεταξύ ευρωπαϊκών και ασιατικών χωρών. Νομίζω ε, ότι αυτό σε έναν βαθμό αποτελεί και ένα πλεξούσιο για τις ε, από τις αναπτυσσόμενες αναπτυγμένες χώρες. Επίσης, αναφερθήκαμε στο ότι μπορούν να υπάρξουν και πολλές ευκαιρίες για την εμπλοκή του ιδιωτικού τομέα. Ένα από τα θέματα που ανέφεραν οι Φιλανδοί συνάδελφοι ε, ήταν το εξή. Αναρωτήθηκαν για την αποτελεσματικότητα του πώς μπορούμε να μειώσουμε τις εκπομπές. Αναφέρθηκαν ε, στις ε, τρεις εναλλακτικέ ε, και μεταξύ των απαντήσεων που θα λάβουμε από τις αναπτυσσόμενες χώρες ε, θα αναφερθούμε και σε ένα ε, ειδικό σχέδιο με των εκπομπών που να βασίζεται στις χρήσεις των τεχνολογιών. θα ήθελα να κάνω και ένα τελικό σχόλιο ότι πρέπει οι ευρωπαϊκές χώρες να συνεργαστούν κυρίως ό,τι αφορά τους ωκεανούς. Και κάτι τελευταίο γιατί μου το ζητήσατε, τρία δευτερόλεπτα. Εγώ ε, στην Ιταλία είμαι στην αντιπολίτευση. Επομένως δεν μπορώ να κάνω κάποια δέσμευση ε, για το να δοθούν ε, περαιτέρω κονδύλια στο Ταμείο. Δεν μπορώ να κάνω οποιαδήποτε δέσμευση εξ ονόματος της κυβέρνησης. Δεν θα μπορούσα να το κάνω τόσοι άλλους. Ακόμη και αν ήμουν στην κυβέρνηση όμως ε, θα στείλω το μήνυμα στους συναδέλφου που βρίσκονται στην πλειοψηφία και μάλιστα στην Επιτροπή Εξωτερικών Υποθέσεων στη Γερουσία ότι αυτό αποτελεί μία από τι μεγαλύτερε προτεραιότητε Γιατί υπάρχουν και περαιτέρω επιχειρησιακές ευκαιρίες ε, για τους οικονομικούς φορείς που σχετίζονται με αυτό. Σας ευχαριστούμε πολύ. Το μόνο που μου απομένει είναι να ευχαριστήσω όλους τους συναδέλφους, όλους ε, τους ε, αντιπροσώπους που ήταν εδώ και που συμμετείχαν. Χωρίς τις δικές σας παρεμβάσεις δεν θα είχαμε μια τόσο πλούσια συζήτηση. Θέλω να προσθέσω ότι οι βουλευτές και οι εγκεκραμένοι εθνικοί αντιπρόσωποι ε, καλούνται ε, στο οίκο της Ευρωπαϊκής Ιστορίας ε, θα έχουμε εκεί και ένα δείπνο σε μπουφέ πριν όμως έχουμε ένα τουρ ουσιαστικά είναι το κτίριο 5 λεπτά απόσταση από το κτίριο του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Και να σας ε, υπενθυμίσω ότι είμαστε το πάνελ 1 και το feedback θα λάβει χώρα αύριο από τις 10 παρατέταρτο μέχρι τις 10.30 εδώ σε αυτή την αίθουσα. Σας ευχαριστώ και καλό σας βράδυ. Υπότιτλοι AUTHORWAVE